Uh, dear colleagues, uh, good morning. I would like to start the meeting. Uh, I would like to... Να ξεκινήσουμε τις εργασίες μας. Καλώς ήρθατε όλες και όλοι. Για το πρώτο σημείο της μέσης διάταξης θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι ο συνήθως αυτή η συνεδρίαση μεταδίδεται ζωντανά. Λοιπόν, Έγκριση τη μέση διάταξη Λάβατε στι 21 Σεπτεμβρίου την τελική εκδοχή τη Μέση διάταξη Δεν έχει ε, εκφράσει κανεί αντίρρηση, ούτε τώρα φαντάζομαι υπάρχει αντίρρηση, οπότε εγκρίνουμε την Μέση διάταξη. Σημείο 2. Ανακοινώσει ε, του Προέδρου, της Προέδρου. Πρώτα απ' όλα να σα ενημερώσω για τι συναντήσει που είχα στα πλαίσια του Brexit μετά την τελευταία συνάντηση τη Επιτροπή ΑΦΚΟ. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι ήμασταν, υπήρξε έντονη δραστηριότητα το τελευταίο διάστημα σε ό,τι αφορά τη διευθύνουσα ομάδα για το Brexit. Έγιναν 5-6 συνεδριάσεις μετά την τελευταία συνάντηση ε, της ε, Κοινοβουλευτικής μας Επιτροπής. Στις τελευταίες συναντήσεις ε, μας απασχόλησε η προπαρασκευή του ψηφίσματος για το Brexit, ψήφισμα που θα υποβάλει στο Στρασβούργο την Τετάρτη, την ερχόμενη Τετάρτη στην Ολομέλεια η Επιτροπή μας. Ε, αυτό το ψήφισμα θα εγκριθεί σήμερα από τη Διάσκεψη των Προέδρων και θα ξεκινήσει στη συνέχεια διαδικασία για την έγκρισή της και στην Ολομέλεια. Δεν έχει ακόμα δημοσιοποιηθεί το ψήφισμα. Να σας πω όμως ότι αναφέρεται σε αυτήν την δέσμευση, την ευρωπαϊκή δέσμευση, να προχωρήσουμε στις διαπραγματεύσεις, να περάσουμε στην δεύτερη φάση το πλαίσιο για το μέλλον καθώς και τα στοιχεία που έχουν να κάνουν με, τη μεταβατική περίοδο. Βεβαίως για να συμβούν όλα αυτά θα πρέπει να σημειωθεί πρώτα στα τρία κεντρικά σημεία, τα δικαιώματα των πολιτών, τα οικονομικά ζητήματα και το θέμα της Βορειοελλανδίας. Μετά τις συζητήσεις ε, χθες το βράδυ στην Διεθνούσα Επιτροπή, ε, στην Διεθνούσα Ομάδα για το Brexit, φτάσαμε στα εξής ε, συμπεράσματα. Έχει συνταχθεί ένα ψήφισμα που ζητά από το Συμβούλιο ε, εφόσον δεν σημειωθεί υπαρκής πρόοδο πρόοδος να ανασταλεί η λήψη της απόφασης ε, για το Δεκέμβριο. Ε, έως τότε θα έχει λάβει η χώρα άλλη μη, άλλο συνεργασιακό διαπραγμάτευση. Γι' αυτό λοιπόν δεν μπορούμε ακόμα να ολοκληρώσουμε τι εργασίε για αυτό το ψήφισμα. Η επόμενη, επόμενο διαπραγματευτικό γύρο ενδέχεται να συνοδευτεί από σημαντική πρόοδο, οπότε δεν μπορούμε να ξέρουμε ακόμα τι θα συμβεί. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για επαρκή ή μη επαρκή πρόοδο τώρα, πριν από το ευρωπαϊκό γύρο. Οπότε, όταν εγκριθεί από τη συζήτηση των Πρόεδρων το σχέδιο ψηφίσματο, θα προχωρήσουμε. Ε, συνάντησα πρόσφατα τον Υπουργό Υπεύθυνο του Πρέσβη στο ΕΒ, συνάντησα και τον Σκοτσέζο Υπουργό τον Μάικλ Ράσελ που ασχολείται με το θέμα αυτό. Συνάντησα λοιπόν εκπροσώπους ε, διαφόρων ε, παραγόντων οικονομικών στην Ευρώπη και το θέμα του Brexit είναι πάντα στην επικαιρότητα. Είχα πει στην ευκαιρία να συναντήσω σε τους συναδέλφους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εμπλέκονται σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Αυτά σε ό,τι αφορά την Επιτροπή ΑΦΚΟ. Εγώ είμαι ανοιχτή σε συζητήσεις ε, ε, και συναντήσεις επ' αυτού. Να σας θυμίσω ότι στις 11 Οκτωβρίου θα λάβει χώρα η ε, Επιτροπή με θέμα το μέλλον της Ευρώπης. Σας ενθαρρύνω να παραστείτε. Θα συμμετάσχει και ο Αντιπρόεδρος Ντομπρόφσκης, ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς ε, και ο πρόεδρος Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Εθνίας που προεδρεύει της Ένωσης αυτή τη στιγμή, ο Μάτι Μάσικας. Και το τέλος θα έρθει και η Μάριν Μαγκίνες, η αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτά στις 11 Οκτωβρίου όλα αυτά. Στη συνέχεια, να σας θυμίσω ότι το τελευταίο διάστημα εργαστήκαμε γύρω από τα έγγραφα για το μέλλον της Ευρώπης ε, της Επιτροπής μας τα έγγραφα εργασίας ε, η γραμματεία εργάστηκε σκληρά ετοιμάζοντας μία ανάλυση για όλους όσους εμπλέκονται ε, στην προπαρασκευή αυτών των εγγράφων ε, ως εισηγητές ή ως ως εισηγητές αυτή η ανάλυση, αυτές οι αναλύσεις έχουν ολοκληρωθεί. Και οι υπεύθυνοι για το καθένα από τα έγγραφα αυτά θα πρέπει τώρα να κάτσουν να σκεφτούν ποια συνέχεια θα δοθεί πάντα βέβαια σε επαφή με την γραμματεία. Ο στόχος είναι να έχουμε οριστικά σχέδια ε, έως τα τέλη Σεπτεμβρίου, δεν μένει πολύ χρόνος. Ε, ελπίζω πάντως να μπορείτε να υποβάλλετε ένα έγγραφο εργασίας εντός του Οκτώβρη ε, ή αρχές Νοέμβρη ενδεχομένως να χρειαστεί να γίνει, λάβει χώρα και έκτακτη συνάντηση της Επιτροπής μας. Θα σας ενημερώσω επίσης ότι θα θυμάστε ότι υπήρχε μια ομάδα εργασία για την αναθεώρηση του κανονισμού το καλοκαίρι ξεκίνησε και η διαδικασία τροποποίησης του ιστορικού κανονισμού και αυτή η ομάδα εργασίας ε, ενεργοποιήθηκε και πάλι, είχε σταματήσει τις εργασίες της μετά την ολοκλήρωση πέρσι. Να σας ενημερώσω λοιπόν ότι η επόμενη συνάντηση αυτή της ομάδας εργασίας θα λάβει χώρα στο Στρασβούργο την 5η το πρωί, 5η 5 Οκτωβρίου, 10 με 11 και μισή. Θα σας τα στείλουμε αυτά θα, μέσω της γραμματείας ε, έγκαιρα. Αυτά για τις ανακοινώσεις της Προέδρου. Και τώρα θα περάσουμε στο σημείο 3, έγκριση των πρακτικών των προηγούμενων συναντήσεων, δηλαδή των συναντήσεων της 11ης Απριλίου, Δευτέρας και 3 Μαΐου. Ε, τα πρακτικά αυτά τα έχετε, εφόσον δεν υπάρχει αντίρρηση έως το τέλος της συνάντησής μας, αυτά τα πρακτικά ε, θεωρείται ότι εγκρίνονται. Θα ήθελα να επιστρέψω την προσοχή σα στο γεγονό ότι στι 10 θα γίνει μια συζήτηση στην διάσκεψη των Προέδρων ε, για το ψήφισμα σχετικά με το Brexit στην οποία θα πρέπει να συμμετάσχω οπότε θα σα εγκαταλείψω ο κύριος Μέσερ Σμιτ θα προεδρεύσει ως αντιπρόεδρος της Επιτροπής ΑΦΚΟ λοιπόν Προτείνω να περάσουμε τώρα στο σημείο 4. Είναι η έκθεση της Mercedes Bresso για την μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ιδίων Πόρων. Θα μας μιλήσει για τις τροπολογίες κτλ. Ε... Ευχαριστώ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως θα θυμόσαστε, είναι μια γνωμοδότηση αυτή για την Επιτροπή Προπολογισμών που επεξεργάζεται το θέμα. Άρα έχουμε κάποια χρονοδιαγράμματα και όρια καθορισμένα. Κατά την άπο... Στη γνωμοδότησή μας αυτή υπευλήθησαν 30 τροπολογίες. Οι περισσότερες από αυτές είναι βελτιωτικές. Διευρύνουν τα διάφορα θέματα, επεκτείνονται στα θέματα που αναφέρουμε, εμπλουτίζουν το κείμενο. Να υπενθυμίσουμε ότι είναι θεσμική η αρμοδιότητα που έχουμε επικεντρώνεται η γνωμοδότηση επιθεσμικών θεμάτων και όχι επί των τεχνικών λεπτομέρειων που αφορούν τους ιδίους πόρους που είναι αρμοδιότητα αυτή άλλων επιτροπών. Δεν διεξήχθη η συνεδρίαση των σκιωδών διότι δεν μπορούσαν να παραστούν οι περισσότεροι. Εργαστήκαμε εχόμενοι σε επαφή μέσω γραμματείας με τα μέλη και καταλήξαμε σε συμβιβαστικέ λύσεις και τροπολογίες που απεστάλησαν στα μέλη. Υπάρχουν συμβιβαστικές λύσεις για τις 30 τροπολογίες. Κάνουμε προτάσεις και περιμένουμε την άποψη των μελών. Για 16 από τις 30 τροπολογίες. Θεωρώ ότι υπάρχει δυνατότητα, θα το δούμε αυτό βέβαια, λέω ότι υπάρχει δυνατότητα να πετύχουμε καλή συμφωνία. Όσον αφορά αυτή τη γνωμοδότηση, βέβαια στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας. Εμπλουτίζοντας το κείμενο και διευκρινίζοντας τις λεπτομέρειες πάντα εντός των αρμοδιοτήτων. Αυτά. Δεν είναι παρόντες και πολύ σκιώδης για να επεκταθώ με η κυρία Μπρέσο. Εκτός μικροφώνη. πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Νταν Πρέντα για το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και την κυρία Μπρέσο. Ε, ήταν ήδη πολύ καλό το κείμενο. Διαπίστωσα ότι έγιναν τροποποιήσεις ε, ε, που βελτιώνουν το κείμενο ούτως ή άλλως καταδεικνύουν την ευρύτερη στήριξη του Κοινοβουλίου ε, στο, στην προσπάθεια που γίνεται για την μεταρρύθμιση του συστήματος ιδίων πόρων ο Ρίτσαρ Κόρμπετ βλέπω ότι συμφωνεί εδώ μαζί μου το σύστημα αυτό δεν είναι ακριβώς παράνομο όπως λέει το αρχικό κείμενο εξαρτάται από, την, από το πώς αντιλαμβάνει το καθένα στους ίδιους πόρους. Τώρα από εκεί και πέρα θα πρέπει να έρθουμε πιο κοντά στο πνεύμα της συνθήκης νομίζω, δηλαδή να αφιερώσουμε ε, περισσότερο χρόνο ε, στους παραδοσιακούς πόρους και να απομακρυνθούμε από τις διαπραγματεύσεις ε, το παιχνίδι των διαπραγματεύσεων για τον δημοσιονομικό προπολογισμό, τον, προπολογισμό της Ένωσης. Τώρα επίσης καλό θα ήταν να βρούμε μια κοινή διατύπωση. Όλοι θέλουμε να ενισχυθεί ο ρόλος του οίκου μας και σε ό,τι αφορά το προπολογισμό της Ένωσης. Ε, θα ήθελα επίσης να χαιρετήσω τη θετική προσέγγιση πολλών τροπολογιών για να καταργηθούν ε, τα στοιχεία του προπολογισμού σε σχέση με το Brexit ε, είναι σημαντικό να σκεφτούμε ήδη από τώρα πώς θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε επαρκή πόρους, επαρκή έσοδα, έτσι ώστε οι πολιτικές της Ένωσης να, είναι αποτελεσματικέ και να επιφέρουν μια πραγματική προσθέμενη αξία. Όπως άλλωστε πρότεινα και στην τροπολογία υπαρθμών 20, το λαμβάνοντας υπόψη την τροπολογία 19 που υπέβαλε η συνάδελφος ε, η Ντανούτα Χούμπνερ και την τροπολογία που επέβαλα εγώ, θεωρώ ότι πρέπει να διευρύνουμε τον κατάλογο των αρχών βάσει των οποίων το σύστημα των ιδιών πόρων ε, έχει θεσπιστεί και να εξετάσουμε και το θέμα τη αυξημένη ορατότητα των πολιτικών που έχουν πραγματική προσθέμενη αξία στον προπολογισμό. Διότι ορισμένε φορέ δεν το βλέπουμε αυτό. Δεν υπάρχει διαφάνεια. Να είναι πιο διαφανή λοιπόν ο προπολογισμό, να είναι λιγότερο περίπλοκο αυτή η στόχοι πρέπει να είναι στην καρδιά της προσπάθειάς μας. Τελειώνοντας να πω ότι στην τροπολογία 28 που υπέβαλα, αλλά και στην τροπολογία 27, αναφερόμαστε σε ένα θέμα πολύ κρίσιμο. Η ενότητα, ο ενιαίος χαρακτήρας του προπολογισμού της Ένωσης πρέπει ε, να το διαφυλάξουμε αυτό. Δεν θέλουμε παράλληλους προπολογισμούς και ανταγωνιστικούς θα πρέπει να προσέξουμε πώς δαπανούμε τα δημόσια χρήματα της Ευρώπης. Ε, στο Στρασβούργο ο Ζαν Κλορ Ιούνκερ, αυτό ζήτησε, ζήτησε ενότητα και νομίζω πρέπει να υποστηρίξουμε αυτή την ιδέα να μην ακολουθήσουμε παράλληλες οδούς που ενδέχεται να οδηγήσουν σε μεγαλύτερο κατακριματισμό, ε, σε μεγαλύτερες διαιρέσεις στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Θέλετε να μιλήσετε για το, για το ECR, παρακαλώ. Ναι, είχαμε μια σύντομη συζήτηση επ' αυτού πριν από λίγο καιρό και δεν έχει αλλάξει η απόψη μου. Θέλω πάρα και εγώ να ευχαριστήσω την κυρία Μπρέσο για την πολύ καλή δουλειά τη. Θα ήθελα επίση να πω ότι δεν θεωρούμε ότι αλλάζοντα απλώ το πώ χρηματοδοτείται, η Ένωση θα ε, αλλάξει την άποψη των ε, πολιτών είναι πολύ τεχνικός ο τρόπος λειτουργίας, ε, πολύ τεχνοκρατικός. Αυτό δεν οδηγεί ούτε σε διαφάνεια, ούτε σε... Ε, ε, ε νομιμοποίηση, όποιο και αν είναι η στόχη ε, όταν περνάμε από ένα εθνικό σύστημα σε ένα υπερεθνικό πάντα υπάρχει πρόβλημα. Γι' αυτό λοιπόν εμείς δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε αυτές τις αλλαγές που αναπόφευκτα θα οδηγήσουν σε απόλυτα κυριαρχία για τα κράτη-μέλη, Προχωρούμε λοιπόν θετικό πνεύμα. Γνωρίζουμε βεβαίω ότι ενδέχεται να μειοψηφίσουμε, αλλά αναμένουμε λοιπόν για τη συζήτηση και τη συνεργασία στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ο Γιάσεν Κοσλίμοβιτ ε, για την Άλντε, την ομάδα Άλντε, να ευχαριστήσω την κυρία Μπρέσο για την πολύ καλή έκθεση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, νομίζω ότι θα είναι αρκετά απλά και εύκολα τα πράγματα παρά τι ιδεολογικέ διαφορέ μα. Ε, επ' αυτού νομίζω ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Όπω είπε ήδη η κυρία Μπρέσο, πρόκειται για μια ε, θεσμική, ε, συνταγματική γνώμη και εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε. Και ένα από αυτά τα θέματα που μα απασχολήσουν είναι το εξής. Όταν θα φύγουν οι Βρετανοί και θα φύγουν, ό,τι και αν σημαίνει αυτό θα φύγουν, ό,τι και αν σημαίνει το Brexit και όποια και είναι τη μελλοντική μας σχέση, αυτό θα οδηγήσει σε απώλεια εσόδων για την Ένωση. Αυτό είναι βέβαιο. Και αυτό θα δημιουργήσει προβλήματα στην Ένωση. Διότι όπως γνωρίζετε, κάποιες ε, κυβερνήσεις ε, αυτή τη στιγμή κάνουν ευθρατεία κατά της Ένωσης. Εμείς τους απευθύνουμε κριτικές και δεν τους νοιάζει. Ε, δέχονται τις κριτικές μας επειδή ξέρουν ότι παίρνουν χρήματα. Τι θα γίνει όμως όταν θα είναι λιγότερα τα χρήματα. Θα δέχονται τις κριτικές μας. Θα συνεχίσουν να συμμετέχουν. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το αναφέρουμε σε αυτή την έκθεση. Επίσης συμφωνώ απολύτως με την ιδέα ότι ο προπολογισμό πρέπει να ψηφιστεί όχι ομόφωνα στο Συμβούλιο διότι είναι ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο ο προπολογισμό έτσι, ε, ένα ευχολόγιο. Το ξέρουμε και σε εθνικό επίπεδο. Σε εθνικό επίπεδο όμω είναι εύκολο. Υπάρχει ένα υπουργό οικονομικών ο οποίο στο τέλο λέει: Ακούστε να δείτε, εντάξει, ε, α, θα κάνω κάποιε επιλογέ. Έχουμε προτεραιότητε. Στην Ένωση είναι πολύ πιο δύσκολο αυτό. Και μπαίνουμε σε ένα παιχνίδι που δεν έχει τελειωμό. Θα πρέπει λοιπόν να ακολουθηθεί η τακτική νομοθετική διαδικασία για την έγκριση του προπολογισμού. Επίσης πρέπει να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία του Brexit για να επανεξετάσουμε το σύστημα ε, διορθώσεων και αποζημιώσεων που χρεούμε σε κάποια κράτη-μέλη. Μία από αυτές τι χώρε είναι δικιά μου, ξέρω γιατί μιλάω, αλλά μιλάμε για ένα σύστημα το οποίο δεν είναι, δεν είναι δεν το καταλαβαίνω καν εγώ. Δεν ξέρω ποιο παίρνει τι, ε, ποιο λαμβάνει υποσμίωση, γιατί. Ε, δεν βγάζει νόημα. Τρίτον, βεβαίως ε, θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη ορατότητα των προγραμμάτων και δράσεων. Έχουμε υποβάλει τροπολογίε σχετικές. Ε, ο προπολογισμό πρέπει να έχει ένα σύστημα δικών του ίδιων πόρων. Ε, από το σύστημα εμπορίας εκπομπών, παραδείγματος χάρη, δεν ξέρω από πού, και πρέπει επίση να αποτυπώνει οι προτεραιότητε. Να πω όμω κάτι εδώ προσωπικό. Τη μισή μου ζωή την έζησα στην πρώην Ιγκοσλαβία και την άλλη μισή στη Σουηδία. Στην πρώην Ιγκοσλαβία όλες οι δημοκρατίες που ανήκαν στη Ιγκοσλαβία πάντα ζητούσαν κάτι παραπάνω. Έλεγαν ότι υπάρχει, ότι αδικούνται. Οι Σλοβαίνοι έλεγαν ότι πληρώνουν περισσότερα από ό,τι πρέπει, το ίδιο και οι Κροάτες. Οι Σέρβοι έλεγαν ναι, εμείς πληρώνουμε μεγάλο το κοσφοπέδιο, αλλά το κοσφοπέδιο είναι ανεξάρτητο, ε, χρησιμοποιούν τις ε, εγκαταστάσεις μας. Ε, ήταν μια ε, συζήτηση χωρίς τελειωμό και αυτό δεν οδήγησε βέβαια στην διάλυση της Ιουγκοσλαβίας, αλλά βοήθησε στις τελευταίες κρίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση βλέπουμε τις ίδιες συζητήσεις. Τις άκουσα. Τις χώρες που λένε ότι «Ναι, εμείς πληρώνουμε για τους Έλληνες ε, που σπαταλούν χρήματα. Οι Έλληνες λένε έχετε τις τράπεζές σας ε, εδώ ε, που μας εκμεταλλεύονται κτλ. Εάν δεν βρούμε ένα σύστημα το οποίο να αποπνέει μια κάποια ισοτιμία, δικαιοσύνη, μια κάποια διαφάνεια και μια δυνατότητα να μπορούμε να εξηγήσουμε στους πολίτες ότι αυτά πληρώνουμε, αυτά κερδίζουμε, ε, τότε διακυβεύεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειαζόμαστε ένα διαφανές σύστημα που να μπορούμε να εξηγήσουμε στους πολίτες. Πληρώνουμε αυτό γιατί αποκομίζουμε τα τάδε ωφέλη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό στην έκθεση. Αυτά. Αναμένω με ανεπιμονησία τη συζήτηση με του κοινού συζητητέ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον κύριο Σαλίμοβιτ. Ο Φάμπιο δεν είναι εδώ. Θέλει κάποιο να μιλήσει για την EFTD. Όχι. Άλλο κανεί θέλει το λόγο. Mercedes. Grazie Presidente. Ο κύριος Τάνεμας θα μιλήσει γι' αυτό πρώτα, σου παρακαλώ. Γι' αυτό. Οι δύο γνωμοδότης θα συνδέονται κάπου. Κυρίως όσον αφορά τις αρχές, θα δούμε στην επεξεργασία τους. Ποιες είναι οι διαφορές. Όσον αφορά τις αρχές και το είπε και ο Μέσο Σμιτ. Θα δούμε. On, on the question whether or not these things, these um, federalist uh, uh steps forward. Uh, για να δούμε ποιο προσέγγιση να ακολουθηθεί λοιπόν. Υπάρχει διαφορά μεταξύ φεντεραλιστών και συνομοσπονδιακών που λένε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι βάση συντονισμού και συνεργασίας και όχι ένα ευρύτερο κράτος που σωθείτε να δημιουργήσετε. Θα ξεκαθαριστούν οι θέσεις. Και αυτό το ρόλο θα ακολουθήσω και στην ψηφοφορία. Ευχαριστώ πολύ. Μερσέντες, έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Καταρχάς, θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη, διότι είπα ότι απεστάλλει. Ε, θεωρούσα ότι τις σαν συμβαστικές, αλλά είναι καθοδόν ακόμα θα τις λάβετε σύντομα. Ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Ήθελα να πω στον κύριο Πρέντα ότι απέσυρα τον όρο επιστολή, letter, ε, παρόλο που λέει, λέει ε, στις συνθήκες ότι πρέπει να βασιστούμε στους ιδίους πόρους. Θέλουμε να ακολουθήσουμε το πνεύμα των συνθήκων. Και απέσυρα αυτόν τον όρο. Για τα άλλα σημεία θα δείτε ότι δέχτηκα τροπολογίες, τις δικές σας και άλλων, που υπενθύμησαν τον ενιαίο χαρακτήρα του προπολογισμού. Συμφωνώ με αυτά που είπε ο κύριος Γιούνκερ. Ο προπολογισμό πρέπει να είναι ένας και ενιαίος, να υπάρχει ένα κονδύλι και αν δίνεται ένα κονδύλι για το ευρώ θα αρκεί να ενταχθεί στον προπολογισμό. Δεν χρειάζεται να υπάρχει ξεχωριστό προπολογισμό απαραίτητα. Και στο θέμα που θέσατε, όπως των επιστροφών, αποζημιώσεων κλπ, του rebate, θα δεχτώ σχετικέ τροπολογίες, ούτω ώστε να είναι σαφέστερη η κατάσταση. Πιστεύω ότι η σαφήνεια, η διαφάνεια μπορούν να αυξηθούν αν έχουμε σαφείς ίδιους πόρους που συνδέονται με τις αρμοδιότητες ενώσεως. Κάποιες προτάσεις που ακούσαμε τις τελευταίες ημέρες, όπως του Προέδρου Μακρόν, ήταν ενδιαφέρουσες. Διότι θα μπορούμε ταυτόχρονα να προστατεύσουμε τις αρνητικές συνέπειες της παγκοσμιοποίησης με θετικά στοιχεία θα προστατεύσουμε λοιπόν την Ευρώπη από τα αρνητικά στοιχεία όσον αφορά το περιβάλλον και τις κοινωνικές πτυχές τι ούτω τρόπος μειώνουμε τα αρνητικά της παγκοσμιοποίησης που έχει σίγουρα και θετικά στοιχεία. Θέλουμε να έχουμε σύμφωνη γνώμη και οι Ευρωπαίοι πολίτες διότι θα υπάρχουν αυτά τα μέσα προστασίας της Ευρώπης που θα παρέχουν πόρους χωρίς να προέρχονται οι πόροι από τις τσέπες των πολιτών. Και οι ίδιοι πόροι είναι αρμοδιότητα της Ένωσης. Αν καταφέρουμε να διοργανώσουμε συνεδρίαση των σκιωδών εισηγητών για να συζητήσουμε τις συμβιβαστικέ, αν θεωρήσετε ότι επειδή είστε ικανοποιημένοι ε, δεν θα κάνουμε περισσότερα. Εξαρτάται από τι αντιδράσει σας αυτές που θα στείλετε όσον αφορά τις προτάσεις τροπολογιών. Δεν ήταν διαθέσιμα τα μέλη όπως προανέφερα και δεν οργανώθηκε η συνεδρίαση των σκιωδών τελικά. Ο κ. Μέσος με είπε κάτι. Κοιτάξτε, δεν αληθεύει απόλυτα ότι η τροποποίηση του τρόπου χρημοδοτήσεως δεν αλλάζει το βάρος για τους πολίτες. Ένας τρόπος χρηματοδότησης που συνδέεται πιο στενά με τις αρμοδιότητες της ενώσεως, άρα να μπορεί να ρυθμίσει η Ένωση τη λειτουργία της χρηματοδότησης και του πόρους, είναι κάτι που αποσαφηνεί την κατάσταση για τους Ευρωπαίους πολίτες. Ότι συνδέονται οι πόροι με την προστιθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Προφανώς για εκείνους που πιστεύουν ότι δεν δίνει προστιθέμενη αξία η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν το συζητάμε για αυτούς. Δεν θα συμφωνούν. Για τις τροπολογίες των φιλελευθέρων σας απάντησα εν μέρη. Πιστεύω ότι πρέπει να πλουστευτεί. Ο καθορισμός, η κατάρτιση του προπολογισμού πρέπει να συνδέεται άρρηκτα με τους ιδίους πόρους της ενώσεως και από αυτού πρέπει να κινηθούν οι εργασίες. Για μας, κυρίως οι θεσμικές πτυχές μας ενδιαφέρουν. Θα παρακολουθήσουμε βέβαια και τις εργασίες των αρμοδίων επιτροπών, κυρίως της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Να εξακριβώσουμε τι το τρόπος ότι οι επιλογές που θα γίνουν στην έκθεση θα συνάδουν με τις θεσμικές αρχές που υπερασπιζόμεθα. Έτσι θα γίνει. Προτείνω να αποδεχτούμε επίσης αρκετές τροπολογίες που αναφέρονται στις προτεραιότητες να προσπαθήσουμε να συνδέσουμε στο βαθμό του δυνατού τους πόρους στις με τις προτεραιότητες της Ενώσεως που καθορίζονται και θα καθοριστούν μάλλον στο επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο και στο επόμενα στρατηγικά προγράμματα της Ενώσεως που θα ακολουθήσει η Ευρώπη ε, μέχρι το 2020. θα προσπαθήσω να μην ετοιμάσω πολλές προτεραιότητες στον κατάλογο. Δεν θα γνωρίζουμε ακόμα τις προτεραιότητες της επόμενης περίοδου προγραμματισμού για την Ευρωπαϊκή Ένωση, παρόλο που έχουμε κάποιες απόψεις και ιδέες γι' αυτό. Όσον αφορά τη δικαιοσύνη και τη διαφάνεια, συμφωνώ απολύτως. Είναι περιπλοκότατα αυτά τα ζητήματα. Όσα σχετίζονται με τον προπολογισμό είναι περίπλοκα. Όσοι ασχολούνται με τον προπολογισμό γνωρίζουν πόσο δύσκολο είναι να έχουμε ένα ε, οικονομικό σύστημα και φορολογικό σύστημα ε, διαφανές. Θα κάνουμε προσπάθειες να πετύχουμε κάτι που βέβαια δεν θα είναι ε, τέλειο, θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατόν. Από αυτά που άκουσα, ως επιτοπλίστων, πιστεύω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε επί συμβαστικών ούτως ώστε η γνωμοδότησή μας τελικά να είναι αρκετά στεναρή, ούτως ώστε να εισακουστεί. Ο κύριος Άνεμανς, κοιτάξτε κύριε Άνεμαν, σας είπα ότι αν δεν συμφωνούμε επί των βασικών αρχών, ίσως συμφωνούμε στις οικονομικές συνέπειες. Η έκθεση που αφορά τη δομή του μελλοντικού δημοσιονομικού πλαισίου, του πολίτους δεν ταιριάζουν με αυτά που μας είπε ο κ. Θα το συζητήσουμε αργότερα. Εδώ είμαι, μπορούμε να το συζητήσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Μεσέντες. Να κάνουμε κάτι ίσως που δεν είναι και τόσο εξυπνό για έναν πρόεδρο. Είχαμε πει αρκετά ότι θα συζητήσουμε μέχρι τις 11, οπότε μόνο στο Στασβούργο μπορείτε να ε, συζητήσουμε τους Αλλά έχουμε προχωρήσει πιο γρήγορα. Αν θες μπορούμε να σας δώσουμε και άλλο χρόνο και να ψηφίσουμε τον Νοέμβριο. Έχουν περισσότερα χρονικά περιθώρια. Μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις, όχι απαραίτητα. Μπορούμε να έχουμε περισσότερο χρόνο για να επηρεάσουμε και το έργο τη Επιτροπή Προπολογισμών. Άρα έχουμε προστιθέμενη αξία. Δεν νομίζω χρειαστούμε παραπάνω χρόνο, λέει η συγκεκριά. Σε άλλο θέμα πάμε, λέει η Πρόεδρος που αφορά τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο είναι η γνωμοδότηση του Harold Hannemans. Harold, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως ήδη ανέφερα, έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα. Για να σας παρουσιάσω ένα κείμενο το οποίο θα ήταν αποδεκτό για όλους. Κάτι που δεν ισχύει, έλαβα τροπολογίες και κατανόησα ότι δεν θα είναι εύκολο να βρούμε βάση για συμβιβασμούς. Και ίσως, όπως κα, κατε, καταδεικνύει συζήτηση επί της γνωμοδοτήσης κ. Μπρεσό, δεν θα προσεγγίσουν οι αρχές. Και είναι δύσκολο να καταλήξουμε σε ένα κείμενο κοινό αποδεκτό. Αν δεν υπάρξει βάση, για συμβιβασμό. Θα ήταν λοιπόν καλύτερο να πάμε στην ψηφοφορία. Είναι σαφείς οι θέσεις, οι τροπολογίες ε, να δημιουργήσουν ένα κείμενο συνεκτικό, ένα κείμενο που έχει μια συνέπεια, δεν πρέπει να χαθεί χρόνος. Οι δύο ψηφοφορίες θα μπορούσαν μάλιστα να συνδεθούν και να λάβει χώρα ψηφοφορία ταυτόχρονα όπως άλλωστε συζητούνται σήμερα ταυτόχρονα τα θέματα. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω τον κύριο Ραντζέλ. Θέλει κάποιο άλλο το λόγο από το ΕΛΚ για το θέμα. Όχι. Πολύ ωραία. Παρακαλώ, σοσιαλιστική ομάδα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ ήθελα να εξηγήσω τον κύριο Άνεμανς, στον εισηγητή, το νόημα των τροπολογιών μας. Ε, Βεβαίω ε, είναι προφανές ότι θα υπάρξουν διαφωνίε αλλά να σα εξηγήσω ε, τις τροπολογίες που έχει υποβάλει η Σοδημοκρατική Ομάδα. Η κυρία Μπρέσο, ο κ. Γιολάινεν και εγώ έχουμε υποβάλει ε, μια σειρά από τροπολογίες ό,τι αφορά αυτή την έκθεση, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προσφέρουμε κάποιες τεχνικές συστάσεις αλλά και κάποια πολιτικά ε, σχόλια. Ε, το τεχνικό σημείο έχει να κάνει με την τροπολογία υπαρθμών 10. Εκεί αναφερόμαστε στο γεγονός ότι αν δεχτούμε, όπως λέει ο εισηγητής, ότι το δημοσιονομικό πλαίσιο ε, θα δομείται ανά πενταετία, κάτι το οποίο μας φαίνεται πολύ λογικό, και υπάρχει συνένεση νομίζω ευρύτερα στο Κοινοβούλιο ε, ότι πρέπει ο προϋπολογισμός ε, να ε, προχωράει παράλληλα με τις θητείες του Κοινοβουλίου. Ε, υπάρχουν κάποιες πολιτικές όμως, όπως οι πολιτικές συνοχής της Ένωσης, όπου είναι πολύ πιο περίπλοκα τα πράγματα κατά την εκτέλεση και θα χρειάζονταν, ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και ο κύριος Άνεμανς θα καταλάβει ότι στην έκθεσή μας ε, αναφερόμαστε σε αυτό. Αναφερόμαστε δηλαδή στην ανάγκη κάποιες πολιτικές ε, να προγραμματίζονται για 5 συν 5 χρόνια με ενδιάμεση αξιολόγηση. Βέβαια είναι η τροπολογία παριθμών 10 αυτή η οποία παρουσιάζει ενδιαφέρον κατά τη γνώμη μας. Τώρα τα πολιτικά στοιχεία έχουν να κάνουν με τρεις ιδέες κυρίως. Ε, πρώτα, να υπάρχει ένας αυτόματος χαρακτήρας ε, σε ό,τι αφορά ε, την, σε ό,τι αφορά τον Brexit. Δηλαδή αυτόματα ε, να ε, υπάρχει προσαρμογή του προπολογισμού. Ε, υπάρχουν κάποια στοιχεία εδώ με τα οποία εμεί δεν συμφωνούμε. Εδώ η έκθεση λέει ότι δεν θεωρείται πολύ πιθανό να αυξηθούν οι προπολογισμοί σε αυτό το πλαίσιο μακροπρόθεσμα. Όχι, εμείς δεν συμφωνούμε με αυτή την ιδέα. Εξού λοιπόν και η τροπολογία ε, που έχουμε υποβάλει να διαγραφεί αυτή η φράση. Ούτε δεχόμαστε την ιδέα ότι η ε, έξοδος του Ηνωμένου Βασιλείου θα μειώσει το προπολογισμό για τον επόμενο συνολικό πλαίσιο. Αυτές οι δύο ιδέες ε, δεν νομίζω να υπάρχει λόγος να αναφέρονται στην έκθεσή μας. Το δεύτερο όμως πολιτικό στοιχείο που ήθελα να αναφέρω είναι ότι σε γενικές γραμμές υπάρχει αύξηση των αναγκών, των αναγκών χρηματοδότησης πολιτικών υπερεθνικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι προφανές ότι η διασύνδεση ενεργειακή, η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, τα ζητήματα της μετανάστευσης, για να μην μιλάμε, μιλήσουμε για την, τα ζητήματα ασφάλειας και άμυνας. Όλα αυτά δείχνουν ότι υπάρχει μία ανάγκη οι πολιτικές της Ένωσης να έχουν μια καλύτερη δημοσιονομική υποστήριξη. Ορισμένοι δεν το θέλουν αυτό, το γνωρίζω. Ορισμένοι δεν θέλουν η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνουν περισσότερα πράγματα. Και δέχομαι ότι σε κάποια σημεία ε, θα πρέπει να ε, γίνουμε πιο ισχυροί, αλλά αλλού πρέπει να γίνουμε πιο ισχυροί. Είναι τόσο προφανές αυτό, που μόνο ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να κάνει κάποια πράγματα και αυτό πρέπει να φανεί και σε πολιτικό πέδο και σε δημοσιονομικό. Κλιματική αλλαγή, ενεργειακή διασύνδεση, έλεγχο των συνόρων, ζητήματα μετανάστευση, άμυνα και ασφάλεια, καταπολέμηση τη τρομοκρατία. Ή θα τα κάνουμε μαζί όλα αυτά, ή θα τα κάνει κανεί. Και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μα και σε πέδο εξόδων. Και αυτό δεν το λέει πουθενά η έκθεση. Και να πω και κάτι βεβαίω για την ανάγκη πολιτικών ε, δαπανών ε, ε, βεβαίως υπάρχουν δαπάνες αλλά υπάρχουν και τα έσοδα όταν μιλάμε για δαπάνες θα μιλήσουμε και για έσοδα και φάνηκε και στην προηγούμενη αίτηση της κυρίας Μπρέσο αυτό ε, στη, η δική μας την εισφορά πρέπει να προτείνει το μελλοντικό δημοσιονομικό πλαίσιο να εξετάσει την δυνατότητα νέων πηγών εσόδων στον προβληματισμό της Ένωσης. Παραδείγματος χάρη, και αυτό είναι κάτι το οποίο η ομάδα μας έχει αναφέρει επανελειμμένα στην Επιτροπή ΕΚΟΝ, γιατί τα κέρδη της Κεντρικής Τράπεζας να μην τροφοδοτούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει αρκετά σημαντικά έσοδα και κέρδη. Γιατί τα κρατάει. Γιατί δεν τροφοδοτεί ε, τους λογαριασμούς ε, της Ένωσης. Ε, γιατί, όπως είπε ο πρόεδρος Μακρόν, να υπάρχει ε, ε, μια φορολόγηση ε, των ε, χρηματιστηριακών συναλλαγών που να έχει ευρωπαϊκή χρειά και που να τροφοδοτεί αυτόματα τον προπολογισμό της Ένωσης για μια σειρά από ζητήματα. Ο κύριος Μακρόν νομίζω στην ομιλία του αναφέρθηκε στη, στη μεταναστευτική πολιτική, αλλά θα μπορούσε να αφορά την άμυνα, όπως είπα εγώ νωρίτερα. Ε, υπάρχει μια τροπολογία υπαρθμών 29, κυρία Νέμανς, που αναφέρει στη δυνατότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον υπάρχει ανάγκη να αντιμετωπίσουμε τις νέες ε, οικονομικές ε, υποχρεώσεις μας, ε, να υπάρχουν και τα κατάλληλα κατάλληλες πηγές εσόδων. Αυτές είναι οι τροπολογίες που έχει υποβάλει η ομάδα μας και βεβαίως θα δούμε αν ο κύριος Άνεμανς ε, θα τις αποδεχτεί. Όχι, εμείς πάντως θα τις ε, υποστηρίξουμε. Ε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ λοιπόν για αυτά που είπατε. Κάποιος από τους φιλελευθέρους θέλει να πάρει το λόγο. Όχι. Ουδής άλλος. Ο κύριος Άνεμανς λοιπόν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως θα σημειώσετε στα πλαίσια της κοινοβουλευτική παράδοσης μια συζήτηση για τον προπολογισμό λοιπόν, η τι δομέ αυτου η το δημοσιονομικο πλαισιο δημιουργει πολιτικα ερωτηματικα και καταδεικνυει ποια ειναι τα ρηγματα τα πολιτικα εντό του κοινοβουλιου μπορουμε λοιπον να πουμε οτι η γνωμοδοτηση κυρια Μπρεσό και η δική μου αποτελούν αντικείμενο πολλών τροπολογιών που δείχνουν πολιτικές αποκλίσεις όσον αφορά το μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Σίγουρα θα ήταν αυταπάτη να πιστεύουμε ότι μπορούμε μέσω μεγάλου συμβιβασμού να ξεπεράσουμε τις διαφορές. Εγώ θα προσπαθήσω, θα διαβάσω προσεκτικά όλες τις τροπολογίες που θα καταφτάσουν και θα δω κατά πόσο μια συνεδρίαση των σκιωδών εισηγητών είναι εφικτή για να πετύχουμε συμβιβασμό. Δεν σας κρύβω όμως ότι για μένα δεν θα είναι και τραγικό αν περάσουμε κατευθείαν ή γρήγορα στην ψηφοφορία. Αναπόφευκτα αυτού του είδους τα θέματα δείχνουν τις πολιτικές διαφορές που, που έχουμε μεταξύ μας όσον αφορά το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την ευελιξία σας. Το χρονοδιάγραμμα που πρότεινε η Γραμματεία είναι να ψηφίσουμε 11 Οκτωβρίου και για τα σχόλιά σας κύριε Χάνεμανς θεωρείτε ότι μπορούμε να πετύχουμε κάποιο συμβιβασμό και υπάρχει και χρόνος για συνεργασία με την Επιτροπή Προπολογισμών διότι πρέπει 4 Δεκεμβρίου να παρουσιάσουν σχέδιο εκθέσεως και θα ψηφίσουν 22 Φεβρουαρίου. Υπάρχουν αντιρρήσεις όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα. Εγκρίνεται. Πάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Το σημείο 6 που προβλεπόταν για τις 10. Τέσσερα λεπτά χαλάρωσης, συνεργασίας, κουβεντούλας, ό,τι θέλετε. So, ladies and gentlemen, the break is over. And we will... Γεια σας και πάλι. Θα αρχίσουμε το σημείο 6 στην ημερήσια διάταξη, καθεστώς και χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και πολιτικών ιδρυμάτων. 13 Σεπτεμβρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την πρόταση νέου κανονισμού. Ίσως θυμάστε, ότι πριν από δύο περίπου μήνες είχαμε μια συζήτηση στην ΑΦΚΟ με εκπροσώπους της ε, Γενικής Διεύθυνσης Finance και τώρα έχουμε μαζί μας εκπροσώπους της Κομισιόν και καλώς ήρθατε. Θα δώσω λοιπόν πρώτα το λόγο στον κύριο Σαν και μετά στους σκιώδεις εισηγητές. Οι ομάδες που δεν έχουν σκιώδεις εισηγητές θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν το λόγο εφόσον το επιθυμούν. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καλημέρα σας. Αγαπητά μέλη, όπως γνωρίζετε, ίσως ο πρόεδρος Γιούνκερ στην ε, ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης το Σεπτέμβριο ανακοίνωσε την, ε, την έγκριση του κανονισμού για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων έτσι ώστε να συνεισφέρουν στην ε, ανάπτυξη της δημοκρατίας και της δημοκρατικής νομιμότητας των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων. Σήμερα από την πλευρά της Κομισιόν λοιπόν καλωσορίζουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τον κανονισμό αυτό σε εσά. Οι αλλαγέ που έχει προτείνει η Επιτροπή ανταποκρίνονται στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τις 15 Ιουνίου φέτος και αναφέρατε και εσείς ήδη την ανταλλαγή απόψεων στις 12 Ιουλίου εδώ στην Επιτροπή ΑΦΚΟ η οποία συνεισέφερε σημαντικά στα προ... στις προπαρασκευαστικές μας εργασίες για τον κανονισμό. Όπως είπαμε, προτείνουμε έναν περιορισμένο αριθμό πολύ στοχευμένων τροποποιήσεων, οι οποίες στόχο έχουν να ε, βελτιώσουν τη δημοκρατική νομιμότητα, έτσι ώστε να αντικατοπτρίζουν καλύτερα το Ευρωπαϊκό Εκλογικό Σώμα, να αυξηθεί η διαφάνεια, έτσι ώστε ο κόσμος να ξέρει ποιον ψηφίζει τα πολιτικά κόμματα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα οργάνωσης και αντιμετώπισης διαφόρων προβλημάτων και χρειάζονται την αντίστοιχη χρηματοδότηση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό οι δύο συνομοθέτες να εργαστούν γρήγορα σε αυτήν την πολύ στοχευμένη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία θα θέλαμε να εγκριθεί τον Απρίλιο του 2018, εάν θέλουμε να έχει αυτό κάποιον αντίκτυπο στη χρηματοδότηση των κομμάτων για τις ευρωεκλογές του 2019. Τώρα θα σας αναφέρω εν συντομία τις διάφορες αλλαγές που προτείνουμε στο σχέδιο κανονισμού. Όπως έχουμε αναφέρει και πριν, οι περισσότερες ε, στόχο έχουν να κλείσουν τα παραθυράκια που έχουμε εντοπίσει. Καταρχάς λοιπόν, ε, αναφερόμαστε στην ε, ιδιότητα μέλου σε πολλά κόμματα. και θα έχουν την ε, δυνατότητα πλέον ομάδες ατόμων και όχι μόνο ένα μεμονωμένο άτομο να ανήκει σε ένα πολιτικό κόμμα, να εγγράφεται μέλος. Μετά αναφερόμαστε στο πολιτικό πρόγραμμα, στο λογότυπο του πολιτικού κόμματος και στην προβολή του προφίλ των ε, υποψηφίων. Έπειτα. Στόχο έχουμε να βελτιωθεί η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και αυτό να φανεί στις ευρωεκλογές. Γι' αυτό λοιπόν προτείνουμε να μειωθεί το ποσό που θα διανέμεται εξίσου σε όλα τα κόμματα από το 15% στο 5% και να αυξηθεί επομένως η χρηματοδότηση για τους ευρωβουλευτές. Επίσης, έχουμε επιλέξει να αλλάξουμε την κλίδα κατανομής και τα ανώτατα όρια από έναν ευρωβουλευτή σε τρεις, οι οποίοι ευρωβουλευτές θα είναι επιλέξιμοι για χρηματοδότηση. Αυτό γιατί αυτή η αλλαγή θα έχει μικρό αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή όλα τα ευρωπαϊκά, ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα εκπροσωπούνται από τουλάχιστον τρεις ευρωβουλευτές. Εάν γίνουν λοιπόν περισσότερες αυξήσεις, τότε θα υπάρχουν νομικά ζητήματα και θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων. Γι' αυτό λοιπόν προτείνουμε και εμείς ένα συγκεκριμένο σταθερό ποσό. Μετά γίνονται κάποιες τροποποιήσεις στις απαιτήσει συγχρηματοδότησης για 10% ε, για τα πολιτικά κόμματα και 5% για τα πολιτικά ιδρύματα. Η εμπειρία που έχουμε από κόμματα και ιδρύματα ε, δείχνει ότι είναι πολύ δύσκολο να αυξηθούν τα επίπεδα συγχρηματοδότησης και τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα αυτοργάνωσης. Μετά, προτείνουμε να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι για την καταπολέμηση καταχρήσεων. Και αναφέρομαι στις εγγραφές πολιτικών κομμάτων ή ιδρυμάτων, οι οποίες πρέπει να πληρούν κάποιες προϋποθέσεις, κάποια κριτήρια και οι πληροφορίες που θα παρέχονται θα πρέπει να μην είναι παραπλανητικές. Επίσης, εξετάζουμε πιθανά μέτρα να ε, επιστραφούν κονδύλια από πολιτικά κόμματα και ιδρύματα και από φυσικά πρόσωπα τα οποία ενδεχομένως ε, ευθύνονται για καταχρήσεις κονδυλίων. Τέλος. Ενώ των εκλογών του 2024 προτείνουμε μία αναθεώρηση των κανόνων χρηματοδότησης ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων εγκαίρως, έτσι ώστε να δούμε τις ε, την εφαρμογή και τις βελτιώσεις που μπορούμε να κάνουμε στο μέλλον. Και σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσω πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε να συζητήσω ήδη σήμερα την πρόταση αυτή μαζί σας και να ευχαριστήσω και όλες τις υπηρεσίε του Κοινοβουλίου για τη στήριξή τους κατά την κατάρτιση του σχεδίου κανονισμού. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Γιώχανσεν. Τώρα το λόγο έχουν οι πολιτικές ομάδες. Ε, Ράινερ Βίλαντ για το ΑΛΚ. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καταρχάς, θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες, όλα τα μέλη, την κυρία Λούνατσακ, τη Γραμματεία και την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όλους όσοι εργάστηκαν και συνεισέφεραν σε αυτήν την πρόταση, η οποία είναι πάρα πολύ λεπτομερής, καθώς επίσης και για την συνεισφορά του στην πρόταση αυτή κανονισμού. Να τους ευχαριστήσω επίσης και για, για την γρήγορη πρόταση αυτή. Καλωσορίζουμε λοιπόν την πρόταση της Κομισιόν γιατί αντιμετωπίζει τα σφάλματα και τα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί στην υφιστάμενη νομοθεσία. Και καλωσορίζουμε επίσης και την περιεκτική αναθεώρηση που προτείνεται. Μια αναθεώρηση η οποία δεν ανήκει στα πλαίσια της ε, προβλεπόμενης αναθεώρησης και του ελέγχου του 2019, αλλά πάει πέρα από αυτό. Θέλουμε κατά τη θέσπιση των νέων κανονισμών να διορθώσουμε τα μεγάλα λάθη και τις παραλήψεις που έχουν γίνει. Κινούμενοι πάντα στα πλαίσια του κράτους δικαίου. Οι σημαντικότεροι λόγοι ήδη αναφέρθηκαν, η πολλαπλή ιδιότητα μέλους, είτε σε ένα είτε σε πολλά ευρωπαϊκά κόμματα. Αυτό είναι ένα από τα κυριότερα σημεία που θέλουμε να αντιμετωπίσουμε. Είναι κάπως δημιουργική κατάχρηση, αν θέλετε, της νομοθεσίας. Έπειτα, θεωρούμε πως είναι πάρα πολύ σημαντικό η χρηματοδότηση των κομμάτων να γίνεται με καλύτερο τρόπο. Η Κομισιόν ήδη ανέπτυξε το θέμα αυτό. αντιμετωπίζει και θέματα φορολόγησης και η προσαρμογή των ανώτατων ορίων προς τα κάτω νομίζω πως είναι πάρα πολύ ρεαλιστική και προσαρμόζεται στις ε, τωρινές συνθήκες. Στόχος βέβαια δεν είναι να λαμβάνει περισσότερα χρήματα ένα συγκεκριμένο ή κάποια συγκεκριμένα κόμματα, αλλά να υπάρχουν κατώτατα όρια και να προσαρμόσουμε έτσι τους κανόνες ώστε να υπάρχει δίκαιη κατανομή πόρων. Έχω μία παράκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η προτινόμενη αλλαγή στο άρθρο 3.1β στην με, στη γερμανική μετάφραση, γλωσσικά τουλάχιστον, έτσι όπως το διαβάζω, δεν αποκλείεται με μονομένα κόμματα να είναι μέλη σε ένα ή περισσότερα ευρωπαϊκά κόμματα. Δεν υπάρχει λοιπόν κάποια σαφήνεια σε αυτό το σημείο και θα ήθελα περισσότερε διευκρινήσει. Να πω τώρα ότι εμεί εδώ στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων πρέπει να εργαστούμε πάρα πολύ γρήγορα, γιατί πρέπει να καταστεί δυνατό στο 2018 για το οικονομικό έτος 2019 να γίνουν ήδη κάποιες ε, προκηρύξεις, κάποιοι διαγωνισμοί έτσι ώστε να τεθεί σε ισχύ το συντομότερο δυνατό. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο μπροστά μας, γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να επικεντρωθούμε στις λεπτομέρειες. Να το πω έτσι χοντρά, πρέπει να συγκυρίσουμε το μαγαζάκι μας. και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τον ελάχιστο χρόνο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο έτσι ώστε να μπορέσουμε ήδη να εφαρμόσουμε αυτόν τον κανονισμό για το 2019. Ήδη έχουμε κάποιες ε, άσχημες εμπειρίες από τις ε, προτάσεις για το δικαίωμα ψήφου στις προηγούμενες εκλογές, οι οποίες μας απασχόλησαν πάρα πολύ και δεν ήταν καθόλου εύκολες. Επί της αρχής δηλαδή πρέπει να επικεντρωθούμε στα ουσιώδη πρώτα και μετά να περάσουμε στα επιμέρους, στις λεπτομέρειες. Ε, γι' αυτό λοιπόν ε, σας παροτρύνω να μην κολλήσουμε στις λεπτομέρειες. Γιατί βλέπω ότι σε ορισμένους τομείς που είναι περίπλοκοι και έχουν πολλές επιπτώσεις σε διάφορους τομείς, είμαστε πολύ λεπτομερείς. Στα κόμματα, ας πούμε, ε, εξαιτία ε, διαφόρων κανόνων για την ισότητα των φύλων, υπάρχουν προδιαγραφές για, το, για την αναλογία ανδρών γυναικών στις επιτροπές των διαφόρων κομμάτων. Αυτό είναι το πρώτο και το βασικότερο θέμα το οποίο μας απασχολεί σε θέματα ισότητας και πραγματικά βλέπω ότι εδώ είμαστε πολύ πίσω. Χρειάζεται να υπάρχουν ανεξάρτητοι εκπρόσωποι των κομμάτων, να υπάρχουν μέλη με συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Χρειάζεται να γίνονται μυστικές εκλογές επίσης. Γι' αυτό λοιπόν όλα αυτά τα θέματα χρειάζεται να τα φροντίσουμε. Όχι όμως σε αυτήν εδώ την αξιολόγηση, αλλά σε επόμενο στάδιο. Και χαίρομαι επίσης για το ότι έχουμε καταφέρει να επιτύχουμε αρκετά μεγάλη συνένεση, έτσι ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε, να εργαστούμε γρήγορα, γιατί είναι αναγκαίο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Μπρέσο έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή διότι δέχτηκε τη εισαγωγή ενός δύσκολου διαλόγου. Ήταν δύσκολο στην αρχή. Στη δική μας Επιτροπή εφαινόταν σχεδόν αδύνατο να πετύχουμε απεμπλοκή για ένα νομοθέτημα που τροποποιήθηκε πρόσφατα και δεν λειτουργούσε ακόμα πλήρως. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δέχτηκε καλά τις απαιτήσει που προβάλαμε και όχι μόνο εμείς, αλλά και οι Ευρωπαίοι πολίτες που μας ζήτησαν να εξετάσουμε το θέμα. Το πώς χρησιμοποιούνται σφαλμένα πολλές φορές οι ευρωπαϊκοί πόροι ρωτούσαν πώς είναι δυνατόν να γίνεται αυτό. Ευχαριστώ την Επιτροπή για την ταχύτητα με την οποία κινήθηκε, την ποιότητα της εργασίας και διότι ενετάχθησε στη δέσμη για των μέτρων για δημοκρατία, διότι η σωστή λειτουργία των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων είναι πάρα πολύ σημαντική για τη δημοκρατία και για τη δημιουργία των πραγματικών ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων, που είναι βασικός μας στόχος στόχος που πρέπει να έχουμε σαν πολιτικές δυνάμεις. Αν δεν υπάρχει ισχυρή παρουσία στεναρών και ορατών ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων, δύσκολο να φανταστεί κανείς πώς λειτουργεί μια ευρωπαϊκή δημοκρατία. Επί της ουσίας των προτάσεων, προφανώς θα συνεργαστούμε για την εξέταση των λεπτομεριών, θεωρώ όμως ότι τα ζητήματα που άπτονται της χρηματοδοτήσεως με μεγαλύτερη αναλογία σε σχέση με τον αριθμό των βουλευτών, με τη σταθερή ποσόστοση. Ούτως ώστε να δημιουργηθούν περισσότερα κόμματα και να διαθέτονται περισσότεροι πόροι, εκεί εμπεριέχονται ενδιαφέρουσες προτάσεις. Συμφωνούμε ότι χρειάζεται να επιταχύνουμε τη συζήτηση στον βαθμό του δυνατού για να εφαρμοστούν τα μέτρα αυτά στις επόμενες ευρωεκλογές. Διότι όπως έλεγα, στις ευρωεκλογέ, αν δεν είναι ορατά τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα, δεν θα είναι πραγματικές ευρωπαϊκές εκλογές αυτές που θα διεξαχθούν υποστηρίζουμε την προσέγγιση. Δεν μπορούσαμε να συζητήσουμε εκτενώς το θέμα στις ομάδες. Όσον αφορά την πρώτερη συζήτηση, πρέπει να πω ότι θέλουμε μεγαλύτερη σαφήνεια της σχέσεως μεταξύ Εθνικού Κόμματος και Αθρίσματος Εθνικών Κομμάτων, συνόλου Εθνικών Κομμάτων με τα Ευρωπαϊκά Κόμματα. Το, το σήμα των κομμάτων η σαφήνεια της εκπροσώπησης της ισότητας των φίλων Εκεί δεν συμφωνώ καθόλου με τον συνάδελφο Βίλεντ. Δεν θέλουμε να επιβάλλουμε την ισότητα των φίλων και την ισορροπία των φίλων αλλά να αναφέρεται ρητά, ξεκάθαρα η κατάσταση και θα αξιολογήσει ο ψηφοφόρος. Πιστεύω όμω ότι είναι κάτι σημαντικό. Τα άλλα ζητήματα βέβαια τίθενται που εγγυώνται το δημοκρατικό χαρακτήρα της λειτουργίας της δομής των κομμάτων. Επίσης και η προσωπική ευθύνη. Πιστεύω ότι όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις και η προσωπική ευθύνη σε περιπτώσεις καταχρήσεων θα πρέπει να είναι η σωστή προσέγγιση. Πρέπει να είναι σαφέστατη όμως η σχέση μεταξύ κατάχρησης και ευθύνης του συγκεκριμένου ατόμου. Ο συνάδελφος Βίλαντ λέει ότι στη γερμανική εκδοχή δεν είναι σαφές το θέμα της απαγόρευσης της συμμετοχής σε περισσότερα ευρωπαϊκό κόμματα από πλευρά των μελών του ιδίου εθνικού κόμματος. Πιστεύουμε ότι καλύπτει αρκετά. Ίσως να υπάρχουν προβλήματα στη μετάφραση ή ασαφίας του κειμένου. Θα το ξεκαθαρίσουμε αυτό, διότι είναι σημαντικό. Αυτές είναι οι πρώτες σκέψεις. Συμφωνούμε απολύτως ότι χρειάζεται γρήγορη επεξεργασία. Πλησιάζουμε στο τέλος της θητείας και θα πρέπει να είναι κανόνας η ταχεία εργασία αν θέλουμε να πετύχουμε πράγματα. εκφράζω μία αρχική άποψη. Δεν εκφράζω την άποψη της ομάδας μου, με αυτό που λέω, αλλά όσον αφορά την τροπολογία που αφορά τη δυνατότητα και Ευρωπαίοι πολίτες μέσω μορφωμάτων που θα εξετάσουμε, μέσω αναφορών, μπορούν να επισημαίνουν ε, καταχρήσεις και ατασταλίες μέσω καταγγελιών. Βέβαια, ξεκινήσαμε από μια καταγγελία που πλευρά νομική δεν μπορούσε να προωθηθεί. Αλλά αυτέ οι αποκαλύψει δημιουργούν κάποιε δυσκολίε πολιτικέ. Θα, πρέπει να μπορούν να εκφράσουν δυσαρέσκεια Ευρωπαίοι πολίτε και να ζητήσουν από μια ανεξάρτητη αρχή που κάνει εξακριβώσει και ελέγχου. Και αν πληρούνται οι προποθέσει, να προχωρά μια έρευνα. Πρέπει να υπάρχει ίσω αυτή η δυνατότητα και ίσω πάνω σε αυτό θα υποβάλουμε τροπολογία κατά λοιπά. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό σε αυτή τη δέσμη για τη δημοκρατία να εισαχθεί και αυτή η πτυχή. Και η πρωτοβουλία των πολιτών, των Ευρωπαίων πολιτών, ίσω πρέπει να ληφθεί υπόψη. Διότι στέλνουμε έτσι ένα μήνυμα προ εκείνου στην Ευρώπη που ζητούν περισσότερη διαφάνεια. Μεγαλύτερη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των Ευρωπαίων πολιτών και να συμμορφωθούμε με αυτά που περιμένουν την Ευρωπαϊκή Ένωση πολίτες. Ευχαριστώ. Επόμενο, επόμενη ομάδα, το ECR. Έχουμε 10 λεπτά που απομένουν για αυτό το θέμα. Δεν το λέω να σας περιορίσω. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, 10 λεπτά είναι 10 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι πολύ σύντομος. Ευχαριστώ την Επιτροπή για την παρουσίαση της πληροφορίες. Να πω κάτι θετικό και κάτι αρνητικό. Η ομάδα μου υποστηρίζει ρυθμίσεις που εμποδίζουν τις καταχρήσεις που θα μπορούσαν αυτές να επηρεάσουν τη λειτουργία των πολιτικών κομμάτων στην Ευρώπη ή να γίνουν, ε, να μην λειτουργούν σωστά τα κόμματα, αν λειτουργούν παράνομα. Είμαστε υπέρ κάθε ρυθμίσεως η οποία ε, εξασφαλίζει την ομιμότητα των κομμάτων. Και όσον αφορά τη μεταφορά των πόρων προς τα κόμματα, η αρχή που αναφέρεται φαίνεται πιο αυστηρή έχουμε την εντύπωση ότι πρόκειται περί μεταφορών πόρων που ευνοούν τα μεγάλα πολιτικά κόμματα και αναφέρομαι στο άρθρο 19. Θεωρούμε ότι αντιβαίνει την αρχή του πλουραλισμού όσον αφορά τα κόμματα και αντιβαίνει στον κανόνα της συμμετοχικής δημοκρατίας όσον αφορά το Ευρωκοινοβούλιο. Στο Κοινοβούλιο παρατηρήσαμε πρόσφατα μία τάση ενισχύσεως των μικρών και μεσών κομμάτων, που είναι αντίθετη η προσέγγιση. Νομίζω ότι αυτή η πτυχή είναι αρνητική στην πρόταση που έχει γίνει. Ευχαριστώ και Ζιωσόφσκι. κύριε Σελίμοβιτς, για, τις, για τους Σας ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω καταρχάς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την δουλειά της. Από τις αρχές του Ιουλίου φάνηκε πόσο σημαντικά είναι αυτά που συζητάμε τώρα και πόσο λεπτό είναι το θέμα αυτό. Νομίζω πως όλες οι ομάδες, όλα τα πολιτικά κόμματα είναι κατά της κατάχρησης πόρων. Αυτό δεν χρειάζεται να το πούμε. Νομίζω ότι η πρόταση είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί θα ενισχύσει την ε, δημοκρατία σε συνταγματικό επίπεδο. Σήμερα όταν ψηφίζουν κάποιον, οι πολίτες δεν ξέρουν αν αυτό θα αλλάξει κάτι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και με τον τρόπο αυτό θα είναι πιο απλά τα πράγματα, πιο εύκολο να το δεις. Ιδιαίτερα με τους ε, κύριους υποψήφιους των κομμάτων. Και οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα λοιπόν να ψηφίσουν όχι μόνο εκείνον που θέλουν να τους εκπροσωπήσει στο Κοινοβούλιο, αλλά και εκείνων που θέλουν στην ηγεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και πρέπει να αποφύγουμε την ε, κατάσταση της τελευταίας φοράς. Αν θυμάστε, ασκήθηκε κριτική στον πρώην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί ήταν άγνωστος ε, σχεδόν. Ο Νάιτζελ Φαράς, μάλλον, αν θυμάστε, είχε αυτή την περίφημη ομιλία που του έλεγε «Ποιος είστε» Και ο λόγος αυτής της πρότασης ε, υποψηφίου ήταν ότι το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν αντίθετο σε οποιονδήποτε γνωστό υποψήφιο. Οποιονδήποτε ισχυρό δηλαδή υποψήφιο. Και όταν ήρθε κάποιος άλλος, τότε εξάσκησαν το χείριστο είδος λαϊκισμού και έλεγαν αυτά τα ποιος είστε εσείς κτλ. Και αυτή η πρόταση λοιπόν πιστεύω πως ε, πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση σε αυτό το θέμα. Έχω κάποια σχόλια. Πρώτον, η απαγόρευση στα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα να ορίζουν υποψήφιους στις εθνικές εκλογές και να συμμετέχουν στις, ε, στα προεκλογικά, στις προεκλογικές εξαρτίες δημοψηφισμάτων. Έχω μια ερώτηση αυτή η απαγόρευση ορισμού υποψηφίων σε ευρωεκλογέ και τις εθνικές εκλογές έχει κάποιο νόημα στις μέρες μας. Όταν μάλιστα γίνεται λόγος για κάποια μεταβατική λίστα για το Ευρωκοινοβούλιο, έχει νόημα να υπάρχει αυτή η απαγόρευση. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σκοπό να αναθεωρήσει αυτή την διάταξη. Μετά, Τι δικαιολογεί αυτή την απαγόρευση συμμετοχής σε εθνικά δημοψηφίσματα. Από το, από, το Brexit και έπειτα έγιναν πάρα πολλές μελέτες σύμφωνα με τις οποίες όχι μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και σε άλλες ε, χώρες οι πολίτες δεν γνωρίζουν τι συμβαίνει εδώ. Δεν καταλαβαίνει ο κόσμος πώς ε, δουλεύουμε, περί τίνος πρόκειται, πώς ψήφος τους έχει κάποιο αποτέλεσμα. Γι' αυτό δεν καταλαβαίνω το νόημα αυτής της απαγόρευσης εδώ. Η συμμετοχή των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων θα πρέπει να βοηθά τους πολίτες να καταλάβουν τι σημαίνουν οι ευρωεκλογέ, τι γίνεται, πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και το να τους απαγορεύει κανείς να συμμετέχουν σε αυτό δεν βγάζει νόημα για μένα. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Άντερσον για τους πρασίνους. Ευχαριστώ πολύ την Κομισιόν για την παρουσίασή της. Να ζητήσω συγγνώμη εκ μέρους του κυρίου Τερικάμπρας που δεν μπορούσε να έρθει σήμερα και θα σας διαβάσω το πολύ σύντομο σημείο, σημείωμα με τα σχολιά του. Αγαπητοί συνάδελφοι, η ομάδα μας, η Πράσινη, ανησυχεί για την κατάχρηση των δημόσιων κονδυλίων. Είμαστε υπέρ της ιδέας λήψης μέτρων για να σταματήσει να γίνεται αυτό. Γι' αυτό λοιπόν υπογράψαμε ένα ψήφισμα μαζί με το ΕΛΚ, τους σοσιαλιστές και την ΑΛΔΕ για μια σειρά μέτρων την οποία καλωσορίζουμε. Δυστυχώς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρόταση της συμπεριλαμβάνει πολλά προβληματικά σημεία τα οποία ε, πλήττουν τα βασικά ε, θέματα της δημοκρατίας, μεταξύ άλλων την προστασία των μειονοτήτων. Η πρόταση για μείωση χρηματοδότησης που και μια χρηματοδότηση που θα δίδεται εξίσου στα πολιτικά κόμματα βλάπτει τον πλουραλισμό του Κοινοβουλίου. Επιπλέον η πρόταση αυτή δεν καταφέρνει να λύσει το πρόβλημα της ε, λάθος κατανομής κονδυλίων, αλλά τα κατα... κατακαιρματίζει τα κονδύλια και αυτά διατίθενται σε μικρά κόμματα μη δημοκρατικά κατανάγκη. Πρέπει να μην αφήσουμε να συμβεί αυτό. Και επιτρέψτε μου και ένα προσωπικό σχόλιο. Εγώ δεν είμαι τόσο υπέρ αυτών των κομμάτων όσο ο κύριος Κιτερικάμπρας. Είμαι φυσικά μέλος του Πράσινου Ευρωπαϊκού Κόμματος. Αναρωτιέμαι όμως αν αυτό το φαινόμενο των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων είναι κάτι που χρησιμοποιεί σωστά τα χρήματα των πολιτών. Είναι σαφές ότι γίνονται καταχρήσεις σε κάποια από τα μικρότερα κόμματα και αυτή η κατάχρηση πρέπει να σταματήσει. Ελπίζω λοιπόν να βρούμε μια κατάλληλη λύση. Σας ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ από την EFDD. Θέλει κάποιο λόγο, χαιρούν πάντα μας ένα λεπτό ε, να επαναλάβω αυτό που είπα και νωρίτερα σε προηγούμενες συζητήσεις εμείς είμαστε υπέρ και θα συνεργαστούμε για οποιαδήποτε μείωση ε, των διπλών ε, μελών και των καταχρήσεων εν πάση περιπτώσει αλλά ε, είμαστε κατά των φημών επίσης ε, που λένε ότι αυτή η μεταρρύθμιση θα προσπαθήσει να μειώσει ε, τη χρηματοδότηση των λεγόμενων λαϊκιστικών κομμάτων. Εδώ πραγματικά με λύπη ε, διαπιστώνω ότι ο κ. Γιούνκερ είπε κάποια πράγματα ε, πριν από δύο εβδομάδες μάλιστα με, μάλιστα καταχειροκρατούμενος ε, εάν υπάρχουν παρά, παράγραφοι όπου θα λέμε ότι κόμματα που δεν συνάδουν με τις αξίες ή που αντιτίθενται στην ευρωπαϊκή δομή, στις ευρωπαϊκές αρχές εδώ ουσιαστικά λογοκρίνεται ιδέες, ιδέες για το μέλλον της Ένωσης. Και αυτό βεβαίως δεν μπορεί, δεν έχει θέση σε καμία μεταρρύθμιση. Λοιπόν, είμαι υπέρ τη μείωση βεβαίως τη κατάχρηση των κονδυλίων αυτών για, προσω... για λόγους, αλλά όχι για πολιτικούς λόγους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Τζέιμς έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το έχω πει και στο παρελθόν, θα το παραλάβω. Δεν υποστηρίζω αυτό που προτείνετε. Να σας πω γιατί. Αυτή η πρόταση είναι υπέρ των μεγάλων κομμάτων, των ε, κατεστημένων κομμάτων. Ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι πολίτες αυτή τη στιγμή απορρίπτουν τα μεγάλα παραδοσιακά πολιτικά κόμματα τα οποία ηγεμόνευσαν ε, τα τελευταία χρόνια τους σοσιαλιστές, τους συντηρητικούς, ε, τους φιλελεύθερους και εμφανίζονται νέα κόμματα, νέες πολιτικές κινήσεις. και βεβαίως από ό,τι φαίνεται εδώ γίνεται μια προσπάθεια να εξουδετερώσουμε, να τον ευρωσκεπτικισμό. Το καταλαβαίνω, αλλά δεν βοηθάει. Αυτές οι δυναμικές τις οποίες αναφέρθηκα δεν φαίνεται να γνωρίζονται πουθενά. Δεν φαίνεται να λαμβάνουμε γνώση. Στην Ολλανδία, στη Γαλλία, στη Γερμανία ε, έχει φανεί η αλλαγή ε, της πολιτικής εικόνας. Και εδώ είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Είτε θα συνεχίσουμε να βλέπουμε τη μείωση της συμμετοχής στις εκλογές στις διάφορες χώρες, διότι δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια άλλη εναλλακτική, οπότε δεν ενδιαφέρει ενδιαφέρεται να πάει να ψηφίσει ο άλλος. Και σε εθνικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό βέβαια. Πρέπει λοιπόν να αποτυπώνεται όλη η βεντάλια των επιλογών Ιδάλλως ε, πραγματικά αποτρέπουμε τον κόσμο να έρθει να ψηφίσει. Θα ήταν καλό να υπόψη αυτά. Ξέρω ότι είναι άβολα αυτά που ακούγονται, ξέρω ότι δεν θέλουμε να ακούσουμε τέτοια πράγματα, αλλά πρέπει να τα εξετάσουμε, να τα πούμε κάπου για να εξεταστούν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω κάποιον άλλον να θέλει το λόγο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Παρακαλώ. Ναι, πρώτα απ' όλα σας ευχαριστούμε για αυτή την πρώτη ανταλλαγή απόψεων και σας ευχαριστούμε και για την υποστήριξη κάποιων ιδεών να πω κάποια πράγματα και να αντιδράσω και σε κάποια πράγματα που ακούστηκαν. Πρώτον, το σημείο αφετηρίας για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ότι εμείς υποστηρίζουμε να έχουμε δυναμικά και ζωντανά πολιτικά κόμματα στην ευρωπαϊκή, σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να συζητούνται τα ευρωπαϊκά ζητήματα ε, είναι ένα στόχο τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής εδώ και πολύ καιρό. Ο μόνος περιορισμός που βλέπουμε εμεί είναι ότι βεβαίως όλοι συμμεριζόμαστε τι αξίες επί των οποίων οικοδομήθηκε η Ευρώπη και αναφέρονται στις συνθήκε αυτές οι αρχές ε, στο άρθρο 2. Αυτό είναι ο μόνο όρο. ο, μόνο, περιορισμό. Αναφερθήκατε στους πολίτες και τη συμμετοχή τους στην πολιτική ζωή. Πρέπει όλοι να συνεργαστούμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται. Ε, ε, ξέρουμε ότι αυτή η Επιτροπή εδώ ε, προσπαθεί να εμπλέξει τους πολίτες στο διάλογο, να τους συμπεριλάβει. Όταν ξεκίνησε η διαδικασία συζήτησης για το μέλλον της Ευρώπης είχαμε πάνω από 2.000 δημόσιες εκδηλώσεις με τους πολίτες που οργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με τις ευρωεκλογέ του 2019 ε, εμείς θα αντιδικοποιήσουμε τις προσπάθειές μας ε, έτσι ώστε οι πολίτες να συμμετάσχουν. Σε ό,τι αφορά τώρα την πρότασή μας νομίζω ότι είναι κοινή η προσέγγιση είναι διτή έχουμε εστιασμένους ε, ε, εστιασμένες αλλαγές που θέλουμε να θέσουμε σε ισχύ πριν από τις αρχές του 2019 για να μπορούν να εφαρμοστούν ενώπιση των επόμενων εκλογών. Ε, Βεβαίω δεσμευόμαστε από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπή να συνεχίσουμε τη στενή συνεργασία μα με τους Ευρωβουλευτέ και τις υπηρεσίε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να συζητήσουμε και άλλα ζητήματα. Ας επικεντρωθούμε όμως σε αυτές τις εστιασμένες τροποποιήσεις αυτή τη στιγμή για τα ζητήματα χρηματοδότηση Πολλοί από εσά αναφερθήκατε στο θέμα αυτό. Το σημείο φετηρία για μα είναι ότι όλα τα πολιτικά κόμματα πρέπει να έχουν τα μέσα για να οργανωθούν. Και σα καλώ να δείτε το σύνολο της πρότασή μας. Πρώτα απ' όλα μειώνουμε ε, την, ε, το τι λαμβάνει το κάθε κόμμα, αλλά αυτό γίνεται αναλογικά. Επίσης ε, μειώνεται και το επίπεδο της χρηματοδότησης. Και αυτό βεβαίως ε, απελευθερώνει πόρους για τα πολιτικά κόμματα. Τώρα για το εκτιμόντος 18 και την απαγόρευση συμμετοχής ε, το να συμπεριληφθούν υποψήφιοι εν δεν το ακουμπήσαμε αυτό στον κανονισμό, γιατί θέλαμε, όπω είπα προηγουμένω, να έχουμε εστιασμένε μόνο τροποποιήσει. Ο κ. Βίλαν τώρα αναφέρθηκε στη γερμανική εκδοχή, θα πρέπει να το εξετάσουμε πολύ προσεκτικά, να εξετάσουμε τι μεταφράσεις. Ε, ένα εθνικό κόμμα ε, μπορεί να ε, υποστηρίζεται από μόνο ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα. Και βεβαίως ε, ε, προσβλέπουμε στη συνέχιση του διαλόγου. Εκτός μικροφώνου η Πρόεδρος. Δεν την ακούμε αυτή τη στιγμή. Θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο ο Μάικελ Άνταμ, ο επικεφαλής ε, ε της ε, Γενικής Γραμματείας ε, ε, αυτής της αρχής για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και ιδρύματα, θέλετε το λόγο για λίγο όμως παρακαλώ, διότι ήδη είμαστε πίσω χρονικά. Ευχαριστώ πολύ θα είμαι πολύ σύντομος. Ε, για μας σε πρακτικό επίπεδο, στο επίπεδο της εφαρμογής, δηλαδή αυτό που εμπεριέχεται στην πρόταση είναι αρκετά προφανές, αρκετά απλό, μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς σημαντικές δυσκολίες. Βεβαίως, ε, εάν υπάρξουν αλλαγές ε, στα κριτήρια αντιπροσώπευσης ε, εκεί στα αυτοτρία. 3 δηλαδή θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορεί να γίνει αυτό μόλις εγκριθεί ο κανονισμός αλλά εν πάση περιπτώσει από διοικητικής πλευράς ε, είναι απολύτως εφικτό αυτό ευχαριστώ ευχαριστώ πολύ να πω ότι ε, ξέρουμε ότι εμείς στην Επιτροπή ΑΦΚΟ ότι εμείς εμείς έχουμε την πρωτοβουλία τώρα θα υποβάλουμε την πρόταση για τους εισηγητές, τον εισηγητή του εισηγητές για αυτό το φάκελο θα εγκριθεί αυτή η πρόταση φαντάζομαι ε, αναμένουμε ακόμα η Ολομέλεια ε, να μας το αναθέσει την ερχόμενη εβδομάδα θα γίνει αυτό καταλαμβανόμαστε ότι επήγει πάντως θέλουμε να ευχαριστήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντως που γρήγορα μας έκανε τη σχετική, μας σχετική πρόταση ε, ανταποκρινόμενη στις προσδοκίες μας Λοιπόν, να κλείσουμε τη συζήτηση εδώ. Όχι, όχι τη συνεδρίαση βέβαια, όχι τη συνεδρίαση, τη, τη συζήτηση για αυτό το θέμα. Ε, Όποιος θέλει να φύγει μπορεί να φύγει βέβαια, αλλά ε, θα γίνει τώρα μια ακρόαση. Η ακρόαση για ένα θέμα το οποίο δεν συζητείται επαρκώς. Δεν είναι αφιερώνεται αρκετός χρόνος. στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αφορά ε, ένα ζήτημα το οποίο το, έχουμε, το μπροστά μας από την αρχή στην ευρωπαϊκή οικοδόμηση ε, οι, οι υποομάδες των κρατών μελών ε, στο Κοινοβούλιο ναι. όποιος φεύγει, φεύγει σιωπηλά εδώ Uh, anybody who wants to talk, please do it. Οπότε παρακαλώ συζητήσεις έξω. Θα ήθελα να ξεκινήσει η ακρόαση για την ε, προέλευση και την ανάπτυξη των υποομάδων των κρατών μελών ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον αντίκτυπο αυτού του φαινόμενου στην ε, ενταξιακή διαδικασία. Έχουμε εδώ τρεις συμπεριγνώμονες για να έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων ο Σαρλ Ντεμασί από το Ίδρυμα Ρόμπερτ Σουμάν, η Αναλένα Κύρχη από το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Εξωτερικών Σχέσεων και ο Ζακ Σίγκερ από το Πανεπιστήμιο της Πάβια. Έχουμε κάπως αργήσει, οπότε τα εισαγωγικά σχόλια θα τα συντομεύσω, ούτως ή άλλως ε, οι παρουσιάσεις είναι που έχουν σημασία. Θα ξεκινήσουμε ευθύ αμέσω και θα δώσω το λόγο Παρακαλώ, μπορεί ο δεύτερος εκεί της σειράς να σταματήσετε να μιλάτε. Δεν αντιλαμβάνεστε πόσο ακούγεστε. Σάλντε Μαρσί, λοιπόν, από το Ίδρυμα Ρόμπερτ Σόμαν πρώτα. Είναι λίγος ο χρόνος, οπότε... Οπότε αν μπορείτε να μιλήσετε 10-12 λεπτά, παρακαλώ. Merci beaucoup, Madame la euh, Ευχαριστώ πολύ και πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να σεβαστώ λοιπόν το δεκάλεπτο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σα. Εν πρώτη, αυτό το θέμα είναι απόλυτα θεμητό και πάρα πολύ επικαιρό. Έτσι δεν περαιτέρω μετά την ομιλία του Πρόεδρου Μακρό με την προοπτική και με την ομιλία για την κατάσταση του ενώσεως που έκανε και ο Γιούγκερ. Το Brexit μας οδηγεί να επανεξετάσουμε την ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως με 27, 33, 34, 35 κράτη αύριο. Ε, βλέπετε ότι έχουμε αύξηση του ευρωσκεπτικισμού, το ξέρετε πάρα πολύ καλά και αναγνωρίζετε και κάτι άλλο που είναι παράδοξο ότι όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις, η μετανάστευση, η αλλαγή του κλίματος κλπ. χρειάζονται συλλογική απάντηση. Και αυτό είναι ενδιαφέρον ότι πρέπει να εξετάσουμε τις διάφορες προοπτικές που υπάρχουν σε υπερεθνικό επίπεδο. Τώρα, συζήτηση για το μέσο Ευρωπαϊκή Ενώση, η διαδικασία τη Πρωτισλάβα που ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του περασμένου έτου, του 2016, και άλλαξε η κατάσταση αν λάβουμε υπόψη τι, είχαμε πέρσι το Σεπτέμβριο με τη φοβία των εκλογών που, επί, που ε, περιμέναμε το 2017. Οι προοπτικέ είναι πιο λαμπρέ σήμερα. Και όπω είπε και ο κ. Γιούκερ, και από πλευρά οικονομική το φως είναι, φαίνεται στην άκρη της σύραγγας. Άλλαξε η κατάσταση και σε διεθνές επίπεδο βέβαια. Έχουμε τη ΣΥΠΑ, τον πρόεδρο Τραμπ και την Κίνα ίσως ε, όσον αφορά τα εμπορικά θέματα. Έχουμε προβλήματα για το κλίμα κλπ. Όλα αυτά και το θέμα των υπομάδων κρατών είναι πιο επίκαιρα στα θέματα. Δηλαδή για να προχωρήσει το καράβι πρέπει να βρεθεί μια λύση. Να προχωρήσουμε μαζί προς τον ίδιο στόχο, έχουμε, το θέμα. έχουμε την εντύπωση ότι όλοι δεν ε, είναι στο ίδιο καράβι προς το ίδιο λιμάνι που κινούμαστε. Μετά θέλουμε να δούμε τη διαδικασία που ακολουθείται για τις προτάσεις και τις εκθέσεις που υποβάλλει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βλέπουμε το Ευρωκοινοβούλιο ε, επίση υποβάλλει τι εκθέσει και καταδεικνύουν όλα αυτά ότι ίσω υπάρχουν όρια και ότι στι 28 δεν λειτουργήσαμε όπω κάναμε σαν 15 μέλη και ίσω 33, 34, 35 χώρε δεν μπορεί να κινηθούν με τον ίδιο τρόπο. Παράλληλα και είναι ένα πρόβλημα που ίσω κάποια κράτη-μέλη αντιμετωπίζουν. Διαπιστώνουμε τον κίνδυνο που υπάρχει αντιστάθμισης ε, διαχωρισμού και προσέγγισης. Όταν έχουμε δύο Ευρώπες ε, ε, μεταβλητής γεωμετρίας, δύο ταχυτήτων, με ομό και τους κύκλους κλπ. Ανακάρτ κλπ. Υπάρχουν, βλέπουμε ότι υπάρχει μια θεωρούν ότι η προσέγγιση μπορεί να διαφοροποιημένη. Έχουν, υπάρχουν τρία οράματα διαφοροποίηση σε εθνικό επίπεδο. Πρώτα απ' όλα, οι Αγγλοσάξονε κάνουν τη διαφοροποίηση, δηλαδή ότι υπάρχει ομοσπονδιακό μένουν εκτό αυτή και επιτρέπεται σε κάθε χώρα που θέλει να μην συμμετέχει όσον αφορά την ολοκλήρωση σε ένα συγκεκριμένο θέμα. Δεύτερο σενάριο, περισσότερο γαλλογερμανικό, διαφοροποίηση μπορεί να δημιουργήσει υποσύνολα που στρέφονται γύρω από το γαλλογερμανικό άξονα και κινούνται προ ολοκλήρωση. Δηλαδή ένωση εντός της ενώσεως δημιουργούνται. Τρίτο σενάριο, κυρίω κεντρική και ανατολική Ευρώπη το ακολουθεί αυτό. Ίσως και συνάδελφο αναφερθεί στη δεύτερη παρέμβαση αυτό. Δηλαδή να ανησυχούν για τα αποτελέσματα που θα μπορούσαν να έχουν οι δύο προηγούμενε προσεγγίσει, διότι οδηγούν σε κατακαιρματισμό τη Ευρώπη. Στην πρώτη περίπτωση και δημιουργούνται κάποιε αποκλειστικέ και στη δεύτερη περίπτωση. Η διαφοροποίηση λοιπόν μπορεί να δημιουργεί κάποιου κινδύνου αν δεν χρησιμοποιηθεί σωστά. Πρώτο κίνδυνο, κατακαιρματισμό υπερβολικό τη διαδικασία τη ολοκλήρωση αυτή καθ' αυτή. Η διαφοροποίηση δημιουργεί ε, θεσμική επιπλοκή παραπάνω στον ε, πολύ συχνά ακούστηκαν επικρίσεων αφορά πώς είναι δύσκολο να αντιληφθούν την όλη κατάσταση ε, οι Ευρωπαίοι πολίτες. Και μπορεί να διαρρεθούν τα κράτη-μέλη όσον αφορά τι τοποθετήσει του και να μένουν κάποιοι εκτό διαφόρων μορφωμάτων και δεν μπορούν να μπουν ή δεν είναι ευπρόσδεκτα να μπουν σε κάποιο μόρφωμα. Οπότε πρέπει να γίνει μια συγκεκριμένη δουλειά. Δεν πρέπει να θεωρήσουμε ότι αυτή η δημιουργία διαφόρων λεσχών ίσω μπορεί να είναι δημιουργία αποκλειστικέ εκθέσει. Πρέπει να υπάρχουν ανοίγματα στις διάφορες κλίμακες, πιστοπαραίτητο αυτό. Στην πράξη λοιπόν, πώς αυτά τα διάφορα επίπεδα μεταφράζονται. Αυτό είναι κάτι που υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, ε, ε, έχει διάφορα επίπεδα με κοινέ δεσμεύσει και από ομάδε κρατών που πιο συγκεκριμένα κινούνται προ μια κατεύθυνση δεδομένη στιγμή. Επιτρέπεται κάτι τέτοιο. Η επόμενη παρέμβαση θα επιτρέψει να υπενθυμίσουμε ότι σε επίπεδο συνθήκων έχει θεσμοθετηθεί αυτή η προσέγγιση. Και βέβαια έχουμε την Ευρωζώνη και τα κράτη, που έχει 19 κράτη μέλη τα 28 και ο χώρος Σέγγεν. Να υποσύνολα. Πολιτικός ισχύει κάτι τέτοιο. Το, το Ίδρυμα Σούμαν ε, δημοσιεύει κάθε εβδομάδα ενημέρωση για την προηγούμενη εβδομάδα στον φάτε επικαιρότητα, τι γίνεται στο Ευρωκοινοβούλιο και τι γίνεται στι διάφορε πρωτεύουσε και τι διάφορου ε, πολιτικού χώρου. Κάθε εβδομάδα λοιπόν έχετε κάποιε πληροφορίε, δύο, τρει, τέσσερι, που δείχνουν ότι υπάρχουν αυτέ οι υποομάδε κρατών. Μπορεί να είναι δύο χώρε, 5, 10, 15, 12. Είναι μια πραγματικότητα ε, που ε, οδηγεί στην ολοκλήρωση στην ευρωπαϊκή διπλωματική προσέγγιση μεταξύ κρατών. Δημιουργείται και μετά δημιουργούνται και πρωτοβουλίες. Πολιτικώς αυτό λειτουργεί ήδη ακόμα αν μπορούμε να πούμε δεν υπάρχει συγκεκριμένο μόρφωμα ενιαίο ε, προνόμιο περισχύ. Η Ευρώπη δεν έχει ομοιογένεια. Ε, είναι μια σύνθεση κοινών συμφερόντων, καμιά φορά αποκλεινόντων ε, στα 28 κάτι μέλη ή καμιά φορά υπάρχει σύγκληση μεταξύ 10, 15, 12. Άρα υπάρχει λογική επιρροών. Δημιουργούνται με γεωμετρική, μεταβλητή γεωμετρία αυτά τα κράτη-μέλη. Κάποια παραδείγματα τα ανέφερε στις μεγάλες ζώνες. Θα αναφέρω και κάποια μορφώματα άλλα, ομάδε κρατών που ακολουθούν ιστορική, η γαλλογερμανική προσέγγιση που ξαναπροωθήθηκε τον Ιανουάριο. Λογικές φόβων, συλλογικών απειλών, όπως εξάρτηση από τρίτε χώρες ε, για το φυσικό αέριο. Οπότε έχετε ομαδοποίηση χωρών οι οποίες έχουν σαν φιλοδοξία να μπορέσουν να κινητοποιηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο όταν βέβαια τα προβλήματα που έχουν τα συμμερίζονται όλα τα κράτη-μέλη. Η λογική των υποδομών, όπω ε, των τριών θαλασσών, σύνο κορυφή των τριών ε, χωρών, είναι οι χώρε Κεντρική Ανατολική Ευρώπη, οι χώρε τη Βαλτική, τη Αδριατική και του Ευξηνού Πόντου και θέλουν να συνεργαστούν σε περιφερειακό επίπεδο, στην επικοινωνία, την ενέργεια, το περιβάλλον. Η τελευταία σύνοδο κορυφή έγινε στι 6 Ιουλίου στην Πολωνία και ήταν ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε ότι υπάρχουν πολιτικοί υπεύθυνοι Κινέζοι και ο πρόεδρο Τρόμπ που εκμεταλλεύτηκαν αυτή την εκδήλωση για να συναντηθούν με κάποια μέρη ε, εκπροσώπου των κρατών. Η λογική διμερή συνεργασία, παραδείγματο χάρη, ο κορυφή αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, υπουργών, ή προέδρων που συναντώνται και μετά υπάρχει το παράδειγμα κατηγορίων των υποκατηγορίων των χωρών, των διαφόρων κρατών μελών, όταν σε κάθε Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάποιε ώρε κατά πολιτική οικογένεια ε, βλέπετε να εμφανίζεται αυτή η μεταβλητή γεωμετρία των πολιτικών σχημάτων, διότι κάθε κυβέρνηση συναρτήσει των εκλογών θα κλείνει προς μια άλλη πλευρά και θα κινηθεί προς μια κατεύθυνση συγκεκριμένη. Και βέβαια έχουμε και πολιτισμική προσέγγιση, πολιτικές αντιλήψεις, ε, όπως είναι η Ευρώπη του Βορρά, κάτι που θα συζητήσουμε μετά, ή λογικές πρόθεσης συλλογικού οράματος και επιρροής, όπως είναι η λογικες προθεσεις του Βίζεγκρατ. Και εκεί ίσως με μεταβλητή γεωμετρία και χωρίς πολιτικές αποχρώσεις και συγκεκριμένες μεροληψίες. Όλα αυτά μεταφράζονται ποικιλοτρόπως. Έχετε λογικές θεσμικές, οι οποίες είναι ιδιαίτερα συγκεκριμένε, πολυμερείς, διμερείς ε, ε, συμφωνίες, opt-out κλπ, συναντήσεις, συμφωνίες που διοργανώνονται από γραμματείες εκδηλώσεις, όπως στην Benelux, ε, μπορεί να είναι ένα κόμμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ένα ευρω... όπως το Συμβούλιο των Σκανδιναβών Υπουργών που αποτελείται από Φιλανδία, Δανία, και από Ισλανδία, Νορβηγία που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως που συμμετέχουν. Οπότε είναι θέμα υποδομών. Υπάρχει και αυτή η δυνατότητα να υπάρχει αυτό το άνοιγμα εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως που μπορεί να οδηγήσει σε μια μορφή ολοκλήρωσης. Λοιπόν, όλα αυτά ε, ακολουθούν μια λογική. Ποια είναι η λογική. Έχουμε μεμονωμένη κίνηση, συλλογική κίνηση που επιβάλλονται ίσως και σε κάποιους άλλους. Για ένα κοινό μέλλον πρέπει να κινηθούμε και πρέπει να διαπιστωθούν διάφορες αποχρώσεις που ανέφερε και ο κύριος Γιούνκερ. χρειάζονται και κάποιοι όροι. Τα ανέφερε και ο μακρόν και ο πρόεδρο Γιούνκερ το είπε. Χρειάζεται, αν θέλουν να προχωρήσουν περισσότερο, να προχωρήσουμε κατά ομάδε των δυνατών πιο μεγάλε και ανοιχτέ. Λοιπόν, διαφρόντα συνεχώ τη φιλοδοξία κάποιων, για το ευρωπαϊκό οικοδόμιο μιλάω, να σεβόμαστε το ρυθμό του καθενό για να πετύχουμε το στόχο, κάνοντα αυτό μπορεί να δημιουργηθεί μια βούληση προόδου που θα είναι υποφελή για όλου. Με κάποια όρια βέβαια. Ίσως αδιαπραγμάτευτε το κράτο δικαίου και αξίε και εσωτερική αγορά. Ακόμα και εκεί ίσω να υπάρχουν ιδιαιτερότητε, αλλά ίσω αυτέ είναι αρχέ που δεν μπορούμε να διαπραγματευτούμε. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Αναλένα Κύρχ για τη δική της παρουσίαση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση και να ευχαριστήσω τον ε, κύριο Μασίν που ήδη μας έδωσε μια γενικότερη εικόνα της ε, κατάστασης, της διαδικασίας τη Λάβα, της ομιλίας του κ. Γιούνκερ για την κατάσταση της Ένωσης, που είναι το πλαίσιο της δικής μου παρουσίασης. Εγώ θα εστιάσω λίγο περισσότερο στις ε, θεσμοθετημένες υπομάδες μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν αποκλειστικά μέλη και θα εστιάσω στο στην συνεργασία των ε, βόρειων χωρών και των χωρών της Βαλτικής. Διότι οι τελευταίες μάλιστα είναι ολοένα και πιο ε, σημαντικές τελευταία. Και τέλος θα αναφέρω και την ομάδα Visegrad και θα αναφερθώ σε κάποιες γενικότερες τάσεις που χαρακτηρίζουν όλες τις ομάδες και τις επιπτώσεις που αυτές έχουν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρουσίασή μου δεν είναι μεγάλη, αλλά όπως ακούσατε και από τον προηγούμενο μιλητή υπάρχει ένα πολύπλοκο σύστημα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα αρχίσω από τις βόρειες χώρες. οι οποίες είναι οι ομάδες χωρών που έχουν την πιο παλιά συνεργασία. Ξεκίνησε με κοινοβουλευτική συνεργασία, το, το Βόρειο Συμβούλιο υπάρχει από το 1952. Η συνεργασία έχει να κάνει με πάρα πολλούς τομείς, από κλίμα, ενέργεια, εκπαίδευση. Υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι του Βόρειου Συμβουλίου στη δεκαετία του 70 όταν ε, δημιουργήθηκε το Συμβούλιο των ε, Υπουργών των Βόρειων Χωρών. Ένα χαρακτηριστικό αυτής της ε, συνεργασίας είναι η εκπεριτροπής προεδρία όπου και υπάρχουν κοινέ κατευθυντήριες γραμμές. Η ομάδα αυτή έχει ένα πολιετές σχέδιο πάνω στο οποίο εργάζεται και αυτό κάνει τη διαφορά ανάμεσα στις άλλες υπομάδες οι οποίες έχουν ε, πιο ε, βραχία συνεργασία. Όπω είπα, το Βόρειο Συμβούλιο ασχολείται κυρίω με θέματα που αφορούν τι βόρειε χώρε. Δεν ασχολείται με την ιδιότητα μέλου Ευρωπαϊκή Ένωση ή με το ΝΑΤΟ, γιατί όταν δημιουργήθηκε το 1952 δεν υπήρχε καν Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν μόνο μια ιδέα η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Αντίθετα, τα κίνητρα για τη συνεργασία ανάμεσα στις βόρειες χώρες ήταν πολύ περισσότερα και ήταν βασισμένα στο ότι αυτές οι χώρες ανήκουν σε μία ε, κοινή γεωγραφικά περιοχή που αντιμετωπίζει τις ίδιες ε, προκλήσεις και έχει τις ίδιες ιδιαιτερότητες η εξωτερική πολιτική και η πολιτική ασφάλεια δεν συμπεριλαμβάνεται παραδοσιακά στη συνεργασία των βόρειων χωρών, ακριβώ γιατί, όπω είπε και ο κύριο Μαρσιλή, υπάρχουν διάφορε υπομάδε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στι ε, βόρειε χώρε έχουμε τη Φιλανδία και τη Σουηδία που, τη, που δεν ανήκουν ε, στο ΝΑΤΟ. Μετά υπάρχουν κάποιες άλλες ε, χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ας πούμε η Νορβηγία και η Ισλανδία. Και μετά η Δανία, η οποία έχει αρκετά opt-out από διάφορες ευρωπαϊκές πολιτικές. Παρ' όλα αυτά, από το 2009 υπάρχει μία επίσημη μορφή συνεργασίας, η Νορντεύκο, που αφορά θέματα άμυνας. Αυτές οι πολλαπλές συμμετοχές σε διάφορες υπομάδες έχουν οδηγήσει λοιπόν ε, στη παραδοσιακή συνεργασία η οποία δεν επηρεάζει τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό όμως έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Στις βόρειες χώρες υπάρχει μια συζήτηση που συνεχίζεται και η παρούσα νορβηγική προεδρία του Βόρειου Συμβουλίου εντόπισε τρεις κύριους τομείς στους οποίους οι χώρες θεωρούν ότι έχουν κοινά συμφέροντα και πως ε, πρέπει να πράξουν με κοινέ αποφάσεις. Δεν υπάρχει κάποιο ε, υπερεθνικό συμφέρον, ε, να πω εδώ, ανάμεσα στις βόρειες χώρες. Η συνεργασία είναι λίγο πολύ αυτόματη. Υπάρχει, λοιπόν, υπάρχουν λοιπόν τομείς της ενέργειας, του κλίματος, του περιβάλλοντος, στις οποίες οι βόρειες χώρες προσπαθούν να εντείνουν τη συνεργασία τους. Τώρα, ήταν κάπως ε, διστακτικές ε, για να αρχίσουν αυτή τη μόρφη της συνεργασίας ε, μέχρι τον Brexit, αλλά αυτό έχει αλλάξει. Υπήρχε ο φόβος δηλαδή, για... υπήρχε ο φόβος μην θεωρηθούν κάποιο μπλοκ χωρών που αποκλείει τις υπόλοιπες. Αυτά όμως τα εμπόδια έχουν ξεπεραστεί και τώρα οι βόρειες χώρες συνεργάζονται και σε αυτά τα θέματα και προσπαθούν να εφαρμόσουν τις αποφάσεις που έχουν ήδη ληφθεί. Τώρα για τις ε, βαλτικές χώρες θα σας παρουσιάσω σύντομα κάποια στοιχεία. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον σύστημα. Είναι μία πολύ καλή περίπτωση υποπεριφερειακής συνεργασίας. Όπως είπε και ο κύριος Μασιλή, εδώ έχουμε από τη μία τις βόρειες χώρες που δεν ανήκουν όλες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. και προσπαθούν να, να ενισχύσουν την συνεργασία τους. Υπάρχει συνεργασία ανάμεσα στις βόρειες χώρες και τις χώρες της Βαλτικής. Υπήρχε βοήθεια με διάφορες αδελφοποίησεις πόλεων κτλ. ανάμεσα στις βόρειες χώρες και σε αυτές της Βαλτικής. Τώρα αυτήν την ε, βοήθεια που τους ε, παρήχαν οι βόρειες χώρες, οι χώρες Βαλτικής προσπαθούν να την παρέχουν με τη σειρά τους οι χώρες της Ανατολικής Γειτονίας. Οι χώρες της Βαλτικής, ακριβώς επειδή είχαν αυτή την πολύ συνεργα... στενή συνεργασία από την αρχή, προσπάθησαν να γίνουν μέλη στα... στο Βόρειο Συμβούλιο. Αυτό δεν έγινε επειδή υπήρχαν ε, αντιρρήσεις από τις βόρειες χώρες. Αλλά υπάρχουν σταθερές σχέσεις ανάμεσα στις δύο ομάδες. Υπάρχει λοιπόν στις χώρες της Βαλτικής μια παρόμοια δομή με εκείνη του, των βορείων χωρών, υπάρχει ένα παρόμοιο συμβούλιο και συνεργασία σε αντίστοιχα επίπεδα. Αυτά σε ό,τι αφορά την σχέση και τη συνεργασία βόρειων χωρών και χωρών της Βαλτικής. Ε, μάλιστα να πω πρόσφατα, να πω ότι πρόσφατα το Συμβούλιο των ε, Βόρειων Χωρών έκανε ένα συμβούλιο για ψηφιακά ζητήματα, το οποίο συμπεριέλαβε και τις χώρες της Βαλτικής. Υπάρχει λοιπόν συνεργασία χωρίς πίεση σε διάφορα θέματα που θεωρούν όλες αυτές οι χώρες ότι τους αφορούν από κοινού. Και υπάρχει επιθυμία για μια μεγαλύτερη ομάδα η οποία θα μπορούσε να ασκήσει ενδεχομένως πίεση σε ευρωπαϊκά θέματα. Τώρα να αναφερθώ και στην ομάδα Βίσεγκραντ, Πολωνία, Ουγγαρία, Τσεχία και Σλοβακία δηλαδή. Αυτή η μορφή συνεργασίας υπάρχει επίσημα από το 1991 και μια μεγάλη διαφορά που πολύ συχνά παραβλέπουμε όταν συζητάμε για το τι μπορούμε να κάνουμε, τι μπορούμε να προγραμματίσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ποιε είναι οι πιθανές άπειλες, είναι ότι αυτή η συνεργασία είναι πολύ λιγότερο θεσμοθετημένη από ότι στην περίπτωση των ευωρίων χωρών και των χωρών της Βαλτικής. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο υπερεθνικό θεσμικό όργανο και η ομάδα Βίσεγκρατ κυρίως έχει στόχο να στηρίξει διάφορα project και την κοινωνία των πολιτών. Υπάρχει δηλαδή συνεργασία η οποία όμως εξαρτάται από την περίπτωση, από την εκάστοτε χώρα που έχει την Προεδρία και από, το, από τη θέληση που υπάρχει για να γίνουν διάφορες ενέργειες. Από τη διάθεση και τη θέληση δηλαδή των εκάστοτε υπουργών, το, των συνθήκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, των συνθήκων που επικρατούν και το πώς βλέπει η υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση τη συνεργασία σε αυτές τις χώρες. Είναι μια σταθερή συνεργασία, δεν υπάρχουν δηλαδή πολυετή προγράμματα. Από την άλλη όμως υπάρχει και αρκετή ορατότητα, γιατί ακριβώς η συνεργασία γίνεται σε επίπεδο υπουργών και ε, πρωθυπουργών και όχι σε τεχνοκρατικό επίπεδο. όπως για παράδειγμα στη συνεργασία των χωρών Μπενελούξ, η οποία είναι πολύ λιγότερο ορατή γιατί εστιάζει συνή, κυρίως σε τεχνικές λεπτομέρειες διασυνοριακής συνεργασίας. Είπαν και κάποιοι πιο πριν ότι αυτό είναι και η προστιθέμενη αξία των ομάδων αυτών, η μη προσκόλληση δηλαδή στη γραφειοκρατία. Βλέπουμε τώρα από την εποχή της κρίσης στην Ουκρανία μέχρι τώρα και από την εποχή που άρχισε να γίνεται συζήτηση για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης πως υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας τις οποίες θα συζητήσουμε αργότερα αλλά και για το μέλλον της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Σλοβακία που συμμετέχει σε όλες τις ευρωπαϊκές πολιτικές είναι μία περίπτωση. Υπάρχουν και άλλες χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή δεν εφαρμόζουν όλες τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Υπάρχουν λοιπόν αυτές οι υποομάδες οι οποίες έχουν περιορισμένη συνεργασία και θα εκτιμούσα πως δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος μία από αυτές τις ομάδες να σχεδιάζει ε, κάτι που θα ε, της παρουσιάσεως ε, ενωμένο μπλοκ. Δεν υπονομεύει δηλαδή τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην περίπτωση της συνεργασίας Μπενελούξ ε, ισχύουν παρόμοια πράγματα. Δεν προλαβαίνω δυστυχώς να τα αναπτύξω. Αλλά αυτές οι ομάδες λοιπόν δεν παρουσιάζονται ως ενωμένες συμπαγείς ομάδες με συγκεκριμένο πρόγραμμα, αλλά υπάρχει ολόνα και περισσότερο η φιλοδοξία αυτές οι ομάδες να θέσουν διάφορους στρατηγικούς στόχους που αποτελούν κοινό συμφέρον για αυτές τις χώρες και να προωθήσουν ε, την κοινή τους, ε, το κοινό τους πρόγραμμα. Δεν προβλέπεται δηλαδή να δημιουργηθεί κάποια υπερεθνική πτυχή σε αυτές τις ομάδες ή να δημιουργηθούν κάποιες πλειοψηφίες σε ψηφοφορίες για διάφορα θέματα. Τώρα πιο συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά τις τάσεις, να σταθώ στα ακόλουθα σημεία. Το δυναμικό που έχουν αυτές οι ομάδες και την κατεύθυνση που θα πάρει αυτή η συνεργασία. Κάτι που πολύ συχνά παραβλέπουμε ε, όχι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στη χώρα μου. Στη Γερμανία παραβλέπουμε αυτές τις υποπεριφέρειες και τα δίκτυα που δημιουργούνται. Υπάρχουν επαφές οι οποίες έχουν σφυριλατηθεί πολλά χρόνια πριν, υπάρχει συνεχής ανταλλαγή πληροφοριών, διαβουλεύσεις πριν από τα Ευρωπαϊκά Συμβούλια. Για παράδειγμα, γίνονται κοινέ αποστολές από αυτές τις χώρες σε τρίτες χώρες, στην Κίνα για παράδειγμα, αλλά και στις Ηνωμένε Πολιτείες. Πολλές από αυτές τις ε, ομάδες λαμβάνουν πρόσκληση από χώρες της Ανατολικής Γειτονίας ή, του, ή στα νότια της Ευρώπης και προσπαθούν να προωθήσουν το πρόγραμμά τους σε διάφορους διεθνείς οργανισμούς. Υπάρχει λοιπόν ε, όλο αυτό το φάσμα των δραστηριοτήτων που δεν είναι και καινούριο. Τώρα, τι προβλέπουμε, ποιο είναι το δυναμικό. Το δυναμικό αυτό έγκυται στα διάφορα έργα υποδομών, στον τομέα των μεταφορών, της ενέργειας και σχετικών τομέων. Οι βόρειες χώρες και οι χώρες της Βαλτικής είναι πολύ μπροστά σε τέτοια θέματα. Έτσι λοιπόν αυτά τα διασυνοριακά προγράμματα έχουν τις τη μεγαλύτερη δυναμική. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι ακριβώς επειδή είναι περιορισμένη η έκταση αυτών των έργων, η μετάδοση του αντικτύπου στις υπόλοιπες χώρες της Ένωσης είναι περιορισμένη. Υπάρχει δυνατότητα βέβαια να αναβαθμιστούν διάφορες υποπεριφερειακές πολιτικές και να γίνουν ευρωπαϊκές, διότι το σκεπτικό πίσω από αυτές είναι παρόμοιο. Μετά, το ίδιο ισχύει και για την αμυντική συνεργασία, που δεν πρόλαβα να αναπτύξω όσο θα ήθελα, αλλά δίδεται έμφαση στη συγκέντρωση πόρων και δυνάμεων σε αυτές τις υποομάδες. Μέχρι στιγμής είναι πολύ μικρό το δυναμικό τους, ε, ασχολούνται κυρίως με θέματα ε, κρατικών προμηθειών, δημόσιων συμφάσεων. Υπάρχουν βέβαια διάφορες ανησυχίες από αυτές τις χώρες που δεν θέλουν να ε, δώσουν κομμάτι της εθνικής τους ε, κυριαρχίας ε, στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Τσίλερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ θα αναφερθώ σε τρία σημεία στην παρουσίασή μου. Πρώτα απ' όλα το θέμα της συμβατότητας επί της αρχής με το δίκαιο της Ένωσης ε, η, η δημιουργία και η λειτουργία των υπομάτων τι είναι αυτό που περιορίζει η δράση των υπομάτων και οι δυνατότητες όταν υπάρχει παραβίαση του δικαίου της Ένωσης. Σε ό,τι αφορά το πρώτο αυτό πρέπει να υπογραμμίσουμε πρώτα απ' όλα και το ανέφερε ήδη ο κ. Μαρσηγή ε, είναι ότι δεν απαγορεύεται η δημιουργία υποομάδων. Το ότι δεν απαγορεύεται δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν όμω όρια. Θα το δούμε αυτό μετά. Σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει και επίσημη αναγνώριση από το δίκαιο της Ένωσης και εδώ πρέπει να ε, πούμε ότι το γεγονός ότι δεν αναγνωρίζεται επισήμως ε, μια υποδομάδα δεν σημαίνει ότι δεν επιτρέπεται. Σε ό,τι αφορά την επίσημη αναγνώριση τώρα, εγώ θα αναφερθώ μόνο στην επίσημη αναγνώριση στο, επίπεδο του πρωτογενούς δικαίου, όχι δηλαδή ε, ε, στις συνθήκες. Δεν θα μιλήσω για συνθήκες μεταξύ κρατών μελών όπως ο, ο, ο μηχανισμός σταθερότητας, θερότες χάρη ευρωπαϊκός, ή το fiscal compact, που δεν είναι ε, πράξεις δικαίου, ε, ούτε η σύμβαση της Σέγγεν, ούτε ε, σύμβαση του ΠΡΙΜ πριν μετατραπεί στη συνέχεια, ούτε συμφωνία μεταξύ Γαλλίας ε, και Γερμανίας των Ηλυσίων, η δήλωση του Βίζεγκρατ που δεν είναι καν ε, νομικός δεσμευτικό κείμενο. Λοιπόν, στις συνθήκες υπάρχει μια επίσημη αναγνώριση της ύπαρξης υποομάδων κρατών μελών. Βεβαίως ε, υπάρχουν υποομάδες ε, για την λειτουργία των θεσμών. Μην το ξεχνάμε αυτό. Ε, ξέρουμε ότι υπάρχουν ε, οι τρεις χώρες που προεδρεύουν της Ένωσης, το τρίο εμπας των προεδριών, η ύπαρξη μιας ε, μειοψηφίας που να μπορεί να μπλοκάρει μια απόφαση μετά την, στο Συμβασμό των Ιωαννίνων, αλλά υπάρχουν παραδείγματο χάρη και το καταστατικό τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προβλέπει υπό για, την, για τον ορισμό ε, αναπληρωτών διοικητικών ε, διοικητών μάλλον. Ε, υπάρχουν και σε περιφερειακό επίπεδο υποομάδες. Ε, το προβλέπει το άρθρο 350 της συνθήκης βάσει, της, βάσει του οποίου η Οικονομική Ένωση μεταξύ Βελγίου και Λουξεμβούργου και το Μπενελούξ αναγνωρίζονται. Αναγνωρίζονται και θα, θα, θα σας πω και πώς. Επίσης, σε μία δήλωση που έχει προσαρτηθεί στην ε, ε, πράξη προσχώρησης του 1995, αναγνωρίζεται η συμμετοχή της Σουηδίας, της Φιλανδίας και της Νορβηγίας στην ε, βόρεια συνεργασία, όπως, στην οποία βρεθήκαμε προηγουμένως. Επίσης, στην πράξη προσχώρησης της Δανίας, της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου η ένωση, μάλλον το τελωνιακό καθεστώς μεταξύ Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου επίσης αναγνωρίζεται με τα βατικά βέβαια ε, όσο θα εφαρμοζόταν οι κοινοτικοί κανόνες. Να περάσουμε τώρα στην πιο σημαντική διάταξη, το άρθρο 350 της συνθήκης, που δεν έχει αλλάξει ε, από τη συνθήκη της Ρώμης και που αναγνωρίζει τι δύο ενώσει μεταξύ Βελγίου και Λουξεμβούργου και των τριών χωρών, Βελγίου, Λουξεμβούργου και κάτω χωρών, των Μπενελούξ δηλαδή. Αναγνωρίζει λοιπόν αυτή την ένωση και του επιτρέπει, επιτρέπει στις χώρες αυτές να εφαρμόσουν αυτά που ισχύουν στι συμφωνίες αυτέ εφόσον ε, δεν ε, πλήττονται οι ισχύοντε κανόνε. Όσο προχωράει λοιπόν η ένταξη ε, στο, και η ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού δικαίου, όλο και λιγότερο οι περιφερειακέ αυτέ ενώσει μπορούν να ε, προβούν σε συμφωνίες, να πάρουν αποφάσεις που να αποκλίνουν. Τώρα, το θέμα της ε, ε, ενισχυμένης συνεργασίας. Εδώ, για τον Πενελούξ, αναγνωρίζουμε τρεις χώρες που έχουν αυτή τη δυνατότητα. Για τις ενισχυμένες συνεργασίες αναγνωρίζουμε τη δυνατότητα. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες από αυτού. Αυτό που έχει σημασία όμως είναι ότι για αυτούς τους τρεις τύπους ε, ενισχυμένης συνεργασίας υπάρχει ένας ανοιχτός χαρακτήρας πάντα. Το ευρώ, παραδείγματος χάρη. Το ευρώ είναι ενισχυμένη συνεργασία, έτσι δεν το αναφέρουμε ποτέ ως τέτοια, αλλά το ευρώ είναι ανοιχτό σε όλα τα κράτη-μέλη. Όχι μόνο είναι ανοιχτό, είναι και υποχρεωτικό για όλους. Το ξεχνάμε αυτό. Μόνο το Ηνωμένο Βασίλειο και η Δανία εξαιρούνται. Η Σουηδία δεν συμμετέχει επί τη βάση μιας νομικής ε, ενός νομικού έτσι, πολύ ε, αφιλεγόμενου. Τώρα από εκεί πέρα υπάρχουν και ανοιχτέ συνεργασίες ε, που είναι ανοιχτέ σε όλους αλλά δεν είναι υποχρεωτικό. Δεν είναι υποχρεωτικές στις δομημένες ε, ε, μόνιμες συνεργασίες και υπάρχουν και οι συνεργασίες ενισχυμένες τρίτο ένσου που έχουν αρχίσει να αναπτύσσονται. Τώρα υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις που αφορούν κάποια κράτη-μέλη ε, συγκεκριμένα. Οι χώρες που έχουν υπερπόντια διαμερίσματα ή υπερπεριφερειακές περιφέρειες. Υπάρχουν σχετικά άρθρα, ε, υπάρχει η χάρτα για τον Πολωνία και τον Βασίλειο, τέτοιου είδους ε, ε, επιμέρους διατάξεις. Λοιπόν, το γεγονός ότι ε, μια υποομάδα δεν προβλέπεται δεν σημαίνει ότι δεν επιτρέπεται κιόλα. Έχουμε μια, ένα σαφές παράδειγμα πολύ ισχυρό στην ομολογία του δικαστηρίου που ήταν και έκπληξη και που αφορά την συνθήκη που δημιουργεί τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Σας θυμίζω ότι ο η συνθήκη τροποποιήθηκε και προσετέθη ένα, μια παράγραφο στο άρθρο 136 που δεν είχε τέθει σε ισχύ όταν έγινε προσφυγή στο δικαστήριο στάθηκε προδικαστικό δικαίωμα δηλαδή ε, ερώτημα μάλλον από τον κύριο Πρίγκλ ε, και το δικαστήριο βρήκε τρόπο να αποδείξει ότι ακόμα σε την περίπτωση ήταν απολύτω εφικτό ε, τα κράτη-μέλη χωρί το άρθρο 36.3 να προβούν σε μια συνεργασία τέτοιου τύπου, ειδική συνεργασία, όπως το Ευρωπαϊκό Συνεργασμό Σταθερότητας. Υπάρχουν αρκετά ενδιαφέροντα στοιχεία στην ομολογία για τις υποομάδες. Περάμε τώρα στο δεύτερο σημείο. Τι είναι αυτό που περιορίζει τη δράση των υποομάδων κρατών μελών στο πεδίο εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης. Τέσσερις είναι οι αρχές εδώ. Πρώτον, είναι η απαγόρευση των διακρίσεων λόγω της υπηκότητας, λόγω της ηθαγένειας. Αυτή η αρχή υπήρχε πάντα στις ε, συνθήκες της Ένωσης και πρέπει εδώ να υπογραμμίσουμε ότι πρόκειται για μια απαγόρευση σε ό,τι αφορά το πεδίο εφαρμογής της συνθήκης. Να δώσω ένα παράδειγμα. Κάποιοι θα θυμούνται ότι πριν από 15 χρόνια ο καγκελάριος Σρέντερ και ο πρόεδρος Ιράκ είχαν αναφερθεί ε, στην δυνατότητα μιας κοινή ηθαγένειας γαλλογερμανικής. Ε, μήπως αυτό όμως θα αποτελούσε διάκριση. Δεν προχώρησε βέβαια. Αν ήταν να δίνεται αυτόματα ηθαγένεια στους μεν και τους δε, γιατί όχι, δεν υπάρχει απαγόρευση. Εάν είναι να δώσουν το δικαίωμα στους Γερμανούς να ψηφίζουν στις, στις ε, βουλευτικές εκλογές στη Γαλλία, ας πούμε, γιατί όχι. Αλλά Εάν μιλάμε για δικαιώματα ηθαγένειας που συνδέονται με την ελεύθερη κυκλοφορία και την άδεια παραμονή το δικαίωμα παραμονής ε, πολιτών της Ένωσης, εδώ μπαίνουμε σε μια πιο δύσκολη ε, σε ένα πιο δύσκολο πεδίο. Δεν επιτρέπεται στους Γάλλους να δώσουν περισσότερα πλεονεκτήματα στους Γερμανούς από τους Ιταλούς ή τους Πολωνούς και του Ε, υπάρχει επίσης το θέμα του σεβασμού του πρωτογενούς δικαίου και του παράγωγου δικαίου ό,τι έχει να κάνει με την εσωτερική αγορά και ό,τι έχει να κάνει με το χώρο δικαιοσύνης, ελευθερίας και ασφάλειας. Μην ξεχνάμε ότι μία από τις πρώτες πολύ σημαντικές αποφάσεις του δικαστηρίου, η απόφαση Βάντεν του 1963, αφορούσε ακριβώς την εφαρμογή από, τα, τις κάτω χώρες της συνθήκης Μπενελούξ στην αθερωμένη εκδοχή του 1958. Ακόμα και το θέμα του Μπενελούξ βέβαια ε, τελικά δεν αναφέρεται στην απόφαση Υπάρχουν μια σειρά από αποφάσεις του δικαστηρίου που έχουν θεσπίσει ουσιαστικά μια αρχή. Το άρθρο 233 τότε, 350 σήμερα, επιτρέπει, επιτρέπεται στα πλαίσια μια υποομάδα όπω τον Πενελούξ να υπάρξει απαρέκκληση από το κοινωνικό δίκαιο εφόσον αυτό του επιτρέπει να πάνε πιο μακριά από το δίκαιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά δεν επιτρέπει βέβαια την θέσπιση διακρίσεων που δεν θα επιτρέπουν την εφαρμογή του κοινωτικού δικαίου. Και δεν μπαίνω σε λεπτομέρειες εδώ. Τώρα, δεύτερη αρχή, η αρχή της ε, πιστής συνεργασίας. Είναι δύσκολο αυτό να το καθοριστεί έτσι νομικά. Είναι και το πιο σημαντική αρχή τις υπομάδες. Μπορούν οι ομάδες, οι αυτές να συνεργάζονται όπως το θέλουν, εφόσον όμως δεν διακυβεύουν την ε, επίτευξη των στόχων της Ένωσης. Ε, και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να μας προσχολεί κάθε φορά που υπάρχει ενίσχυση συνεργασίας που δεν προβλέπεται από τη συνθήκη, ε, αντίθετα δηλαδή από το Μπενελούξ και την Βελγολουξοβεργανή Ένωση, και κάθε φορά που υπάρχουν συμφωνίες στα πλαίσια της λειτουργίας των θεσμικών οργάνων σε σχέση με αυτή την αρχή της πιστής συνεργασίας υπάρχει σχετική νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και πιο συγκεκριμένα για τον Μπενελούξ. Τρίτη αρχή που συνδέει τα κράτη-μέλη, το μονοπόλιο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να δημιουργήσουν δικαιοδοσίες στις οποίες θα μεταφέρουν, θα προσδώσουν δικαίωμα ε, απόφασης και για υποθέσεις που έχουν να κάνουν με το κοινοτικό δίκαιο. Η Ιρλανδία, παραδείγματος χάρη, έχει υποβάλει ε, στο Διεθνές Δικαστήριο της Θάλασσας ένα ζήτημα που, ε, μια που είχε με το Βασίλειο και υπήρξε προσφυγή. Προσφυγή επί παραλήψη και ε, η οποία κερδίστηκε διότι αφορούσε το κοινοτικό δίκαιο. Μπορούμε να πούμε μάλιστα ότι το Μπενελούξ έχει ένα δικαστήριο που έχει πάρει περίπου 350 αποφάσεις που υπάρχει και αυτό το δικαστήριο αναγνωρίζεται ως ένα δικαστήριο των κρατών μελών για να μπορεί κάποιος εκεί να στείλει μια προδικαστική, ένα προδικαστικό ερώτημα. Ε, κάτι άλλο σε σχέση με άλλους ε, ενώσεις που δεν αναφέρθηκαν. Υπάρχει η Σύμβαση των Άλπαιων που προβλέπει ένα διατητικό δικαστήριο. Η Σύμβαση των Άλπαιων αφορά βεβαίως και στοιχεία του κοινοτικού δικαίου. Αυτό που είναι περίεργο εδώ είναι ότι η ίδια η Ένωση συμμετέχει στη Σύμβαση των Άλπαιων. Εάν δηλαδή τα μέλη της Σύμβασης των Άλπαιων ε, παραβιάσουν το μονοπόλιο ε, του δικαστηρίου, θα πρέπει να παρέμβει η Κομισιόν εις βάρος της ίδιας της Κομισιόν. Λοιπόν, ποιε είναι οι δυνατότητες δράσης όταν υπάρχει παραβίαση του κοινοτικού δικαίου. Το πιο σημαντικό είναι βεβαίως η προσφυγή η διαδικασία επί ε, και επί παραβάση. Ε, σε κάποιες περιπτώσεις αυτό συνέβη απέναντι σε κράτη-μέλη μεταξύ των οποίων του Μπενελούξ. Ε, αυτό που ξεχνάμε είναι ότι υπάρχουν και προδικαστικές, προδικαστικά ερωτήματα και έτσι ακόμα και τα κράτη-μέλη συμφωνούν να μην κάνουν κάτι ένας πολίτης μπορεί να ενεργοποιήσει να, να θέσει ε, να ξεκινήσει μια διαδικασία περιπτώσει προσφυγής. Στην συζήτηση από εκεί πέρα θα δούμε κατά πόσο αυτά τα όρια μπορούν να αυξηθούν ή αν πρέπει να μειωθούν στα πλαίσια μια ενθόρησης συνθήκων. Αυτά ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πάρα πολύ, καθηγητά Τσίλερ. Δίνω το λόγο στους συναδέλφους. Η Περβάμς Περές είναι η πρώτη. Ευχαριστώ για τις παρεμβάσεις. Είναι πολύ ανανεωτικές. Μπορούμε να καλύψουμε όλο το φάσμα. Ενώ εν γέννη ενδιαφερόμεθα με κάποια σημεία τα πλέον ορατά. Αυτή η ακρόαση που έχει προγραμματιστεί προκαιρού εντάσσεται στο πλαίσιο το ιστορικό που γνωρίζουμε. και είναι ακριβώς στην καρδιά των συζητήσεων. Τις ανησυχίες που εξέφρασε η Καγκελά στη Γερμανία, την ομιλία του Ζαν Κλωτιούν για την κατάσταση στην Ένωση και τα όσα είπε και ο πρόεδρος Μακρόν. Από την πλευρά μου, όσον αφορά την Ευρωζώνη, δεν θα σε εκπλήσει ότι μπαίνω ότι ο τρόπος στο θέμα και από αυτή τη γωνία έχει ξεκινήσει μια πολύ ουσιαστική συζήτηση στρατηγικής σημασίας. Πρέπει να χρησιμοποιηθεί σωστά το νομικό προστάσιο για να, κάνουμε τη, να πετύχουμε την πρόοδο που θέλουμε. Πολλοί από εσά αναφερθήκατε στις διατάξεις που συμπεριλαμβάνονται στις συνθήκες. Το άρθρο 350 που είναι η πιο επίσημη μορφή αναγνώρισης υποομάδας, η πιο ολοκληρωμένη μορφή αναγνώρισης είναι αυτή, κανείς δεν αναφέρθηκε όμως στη συζήτηση που διεξήχθη στα πλαίσια της συνέλευσης που αφορούσε το άθρο 250 ήταν ε, πολύ ενδελεχή συζήτηση που διεξήχθη. Είχα αποβάλει και εγώ τροπολογίες εν αυτή τη εννοία για να χρησιμοποιήσουμε αυτό το πλαίσιο σαν πλαίσιο αναφοράς για την Ευρωζώνη. Ο πρόεδρος Ζισκάρ ενδιαφερόταν τα μάλα για αυτή την προσέγγιση. Είμαστε στην Επιτροπή ΑΦΚΟ που είμαστε ανοιχτοί στον αφάσεις προοπτικές. Σημαίνει λοιπόν ότι την ημέρα που θα έρθει αυτή η μέρα και θα ξαναανοίξουμε τις διαπραγματεύσεις για τις συνθήκες θα πρέπει να τροποποιηθεί το άρθρο 350. Θα διευρυνθεί. Η χρήση του θα αυξηθεί. Ή με ήπιο τρόπο, soft τρόπο, να κινηθούμε μέσω ενισχυμένης συνεργασίας ή μέσω διαθρωμένης συνεργασίας ε, και διευρυμένης συνεργασίας να κινηθούμε. Είμαστε νομοθέτες και αυτό είναι το πρώτο χρήσιμο ερώτημα πρέπει να τεθεί. Άλλο ερώτημα. Το επόμενο για τη λειτουργία του, για το, για το σύμφωνο για τα δημοσιονομικά. Αυτό έχει εξαιρεθεί από τις αρμοδιότητές σας. Μπορεί να λυθεί το πρόβλημα. Όμως, τι πρέπει να πει το Κοινοβούλιο έναντι ενός ε, μηχανισμού, ενός νομοθετήματος που δημιουργείται εκτός συνθήκων, δημιουργείται μια αποδομάδα κρατών μελών ακολουθώντας διακυβερνητική προσέγγιση. Καταχρώμενα και εκμεταλλευόμενα τα θεσμικά όργανα της Ενώσεως, δηλαδή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ΔΕΚ. Αυτό δημιουργεί πρόβλημα και πρέπει να συζητηθεί. Τώρα, όσον αφορά τις υπομάδες και το δίκαιο που τα διέπει, θέλουμε να δούμε ποιες συνέπειες υπάρχουν και πώς διαρθρώνονται αυτές. Άλλο ερώτημα. Έχουμε στα δικά μου το μέλλον της Ευρωζώνης. Κανείς από εσά. Και ζητώ συγγνώμη γιατί δεν άκουσα την αρχή της συζήτησης, ίσως το αναφέρατε, όμως για την Επιτροπή μας και το Κοινοβούλιο αυτό που μας απασχολεί επίσης είναι ο, ο δημοκρατικός έλεγχος Πώς διαθρώνετε με τις υποομάδες. Είναι ένα θέμα που μας απασχολεί συνεχώς. Το λύσαμε αυτό. Χρησιμοποιώντας ένα ταμπού. Θα γίνει κρισίμου σημασία στο θέμα. Αντάλλαξα επιστολές με κάποιους πάνω σε αυτό. Μήπως θα φτάσει ο κόμπος στο χτένι όταν δημιουργηθεί μια οντότητα δημοσιονομική. Ποια προσέγγιση θα ακολουθηθεί από το Κοινοβούλιο για το δημοκρατικό έλεγχο μιας υποομάδας σε αυτή την περίπτωση. Δεν το τόνισε ιδιαίτερα αυτό ο κ. Γιούνκερ για προφανείς λόγους. Αν θέλουμε όμως ε, να μπει το Ταμείο Στατικών Επενδύσεων... Ε, euh, euh, τα κράτη-μέλη λοιπόν πρέπει να συμμετέχουμε. Ο μηχανισμός ε, δημοσιονομικής σταθερότητας να ενταχθεί, πώς θα ενταχθεί. Λοιπόν, χρειάζεται να δούμε πώς το βλέπετε εσείς το θέμα. Η συνεισφορά σας μπορεί να είναι πάρα πολύ χρήσιμη όσον αφορά αυτό το θέμα. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους τρεις ομιλητές που παρουσίασαν την όλη προβληματική των υποομάδων, εγώ από την πλευρά μου, από την πλευρά μας. Η ε, κυρία Μπερές το ανέφερε το θέμα και συμμερίζομαι τα ερωτήματά τη όσον αφορά τα θέματα της Ευρωζώνης κλπ. Τι γίνεται με τη δημοκρατία, το δημοκρατικό έλεγχο των υπομάδων. Θα ήθελα να επικεντρωθώ επί μιας υπομάδας που δημιουργεί περισσότερα προβλήματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτή είναι η υπομάδα του Βίζεγκραντ επικεντρώνομαι επ' αυτού του σημείου διότι πιστεύω ότι τη αυτή περίπτωση πρέπει να κινηθούμε πέρα της τεχνικής εξετάσεως της λειτουργίας της υποομάδας που είναι κυρίως υπερεθνικό επίπεδο με προγράμματα πολιετή κλπ. Κατά την άποψή μου φτάνουμε φτάνουμε σε διαφορετική ιστορική μνήμη όσον αφορά αυτή την ε, υπομάδα, ιστορική μνήμη της Ευρώπης, διαφορετική αντίληψη όσον αφορά τις απειλές. Διαφορετική αντίληψη που μπορεί να γίνει κατανοητή, είναι κατανοητή λέγω, διότι κατά κάποιο τρόπο οι χώρες του Βίζεγκραντ είναι ε, το μετερίζει ε, στα όρια, είναι στα όρια της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως ήταν η Γερμανία, η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας παλιά ήταν στα όρια της Ευρώπης. Τώρα έχουμε κινηθεί προς ανατολικά στον φρατόριο. Αυτό όσον αφορά την αντίληψη των απειλών. Αποτέλεσμα της διαφορετικής ιστορικής μνήμης και αντίληψης των απειλών είναι κάτι που δεν συζητήθηκε όταν διαπραγματευόμαστε τη διεύρυνση. Δηλαδή, ποιο είναι το ε, όραμα της κυριαρχίας. Όσον αφορά την κυριαρχία, την εθνική κυριαρχία, υπάρχει βαθιά διέρεση μεταξύ των υποομάδων που αναφέρθηκαν. Ευρωζώνη, ε, ε, οι χώρες της Συμφωνίας της Συμφωνίας και της Βίζεγκραντ. και οι θέσεις και τοποθετήσει των υποομάδων καθορίζεται από την ιστορική μνήμη και τι θεωρείται σαν μόνιμη απειλή και κίνδυνος. Και υπάρχει ο κίνδυνος ε, μέσω της ιστορικής μνήμη να επαναληφθεί η ιστορία. Και υπάρχει και ένα όραμα όσον αφορά τη χάρτα θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρώπη. Πάνω σε αυτό είναι ένα σύνολο αξιών αυτή η χάρτα των δικαιωμάτων και οι αξίες μπορεί να είναι συγκεκριμένοι, διότι οι αξίες είναι κάπως υποκειμενικές. Δεν θεωρείται ότι αποτελούν νομική βάση της Ένωσης. Προδιαγραφές που με τις οποίες συμμορφώνται όλα τα κράτη ακόμα και αν έχουν διαφορετικές ιστορικές μνήμες και παραδόσεις. Άλλος τομέας όπου υπάρχει απόκληση ιστορικών μνημών είναι της συνεργασίας της θεμητής που δεν λειτουργεί όπως με τους πρόσφυγες δεν λειτουργεί σε αυτή η συνεργασία για τις μετεγκαταστάσεις, τις ποσοστώσεις μετεγκαταστάσεων των προσφύγων. Το όραμα διέφερε. θεωρήθηκε ότι δεν παραλαμβάνονται αποφάσεις για αυτό το θέμα σε επίπεδο νόσους διότι αυτό είναι κυρίαρχο δικαίωμα ε, των χωρών. Και είχαν διαφορετική άποψη οι χώρες Βίζεγκραντ. Αυτά τα θέματα πρέπει να τα συζητήσουμε. Δεν ξέρω αν υπάρχουν εκπρόσωποι των χωρών Βίζεγκραντ παρόντες εδώ. Όμως είναι ένα θέμα που θα μας συνοδεύσει τα επόμενα έτη και θα γίνεται όλο και πιο σημαντικό. Ευχαριστώ. Uh, thank you very much. Ευχαριστώ πολύ, Μπάρμπαρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να συγχαρώ του τρει Όλα αυτά τα οποία μα εξήγησαν θα τα εξετάσουμε βεβαίω, θα τα μελετήσουμε και θα μα χρησιμεύσουν ιδιαίτερα για να συνεχίζουμε να δημορφώνουμε πολιτικές απόψεις, διότι ε, και θέλω να συμφωνήσω με τις προηγούμενες ομιλήτρες, διότι και τα δύο θέματα τα οποία έθεσαν είναι εξαιρετικά σημαντικά και θα πρέπει να τα συζητήσουμε όλα αυτά πολύ περισσότερο, πολύ πιο έντονα στο μέλλον. Χρειαζόμαστε λοιπόν την τεχνική υποστήριξη που μας ε, δώσατε. Υπάρχει ένα ζήτημα που με απασχολεί ιδιαίτερος. Ένα πολιτικό ζήτημα. Το θέμα της συνοχής, της συνέπειας μεταξύ μιας υποομάδας και του τι είμαστε εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση, τι προβλέπει η συνθήκη και ποια είναι τα στοιχεία ερμηνείας που έχουν να κάνουν με την φιλοσοφία που έχει δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε πολιτικό επίπεδο. Είναι πολύ σημαντικό και αυτά να τα συντάξουμε στη συζήτηση όλα αυτά που προσπαθούμε να οικοδομήσουμε, όλα αυτά που είμαστε, προέρχεται από τις τάξεις του πολέμου. Προέρχονται από τις επιπτώσεις ενός εθνικισμού τοξικού, από τη δημιουργία της θυματοποίησης κάποιων χωρών απέναντι σε άλλες και από τη δημιουργία ηγεμονιών που αποκλείουν τους υπόλοιπους και αποκλισμούς ελευθερίας ε, πολιτικής συνείδησης όποιος δεν είναι ε, ε, αυτό που πρέπει δεν είναι ο καλός Γερμανός παραδείγματος χάρη έπρεπε να, μην υπάρχει πια να αφανιστεί στη συνέχεια η Ευρωπαϊκή Ένωση και η οικοδόμησή της βασίζεται σε, βασίστηκε σε αυτά τι σημαίνει αυτή τη στιγμή τη κράτη-μέλη και φυσιολογικό είναι αυτό διότι τα κράτη-μέλη έχουν συμφέροντα. Βεβαίως υπόκεινται σε κανόνες, έτσι, στους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν κάποιοι, κάποια συμφέροντα τακτικά, ε, με τα όρια, όχι στις διακρίσεις ε, και βεβαίως ε, πιστή συνεργασία, αναφέρθηκε η κυρία Σπινέλη προηγουμένως. Όμως, όταν αναμοχλεύουμε την ιστορία όταν υπάρχει θεματοποίηση απέναντι στι Βρυξέλλε, όταν δεν υπάρχει πιστή συνεργασία, όταν ψάχνουμε να βρούμε στοιχεία ε, σε μια υποομάδα που το καθιστούν λόμπι ή το καθιστούν περιούσιο, ε, περιούσια υποομάδα, α πούμε, όλα αυτά οδηγούν σε μια απειλή. Κανείς από εμά ε, δεν κατέχει την αλήθεια για το τι είμαστε και το τι οικοδομούμε. Αλλά πρέπει να είμαστε ειλικρινεί. Πρέπει να σκεφτούμε και να αντιμετωπίσουμε αυτά που συμβαίνουν σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να σκεφτούμε και να συζητήσουμε με σαφήνεια και με ειλικρίνεια. Διότι εδώ μπορεί να έχουμε μπροστά μα μια πραγματική απειλή για την Ευρώπη που οικοδομούμε. Και βεβαίω στο Βίζεγκραντ υπάρχουν τέτοιου είδου στοιχεία. Ευχαριστώ, Μάιτε, κυρία Μπρέσο. Ε, ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ τους φιλοξενούμενούς μας για τις παρεμβάσεις τους. Ήταν ισορροπημένες οι παρουσιάσεις μας παρουσίασαν άκρως ενδιαφέρουσες προοπτικές και οπτικές γωνίες. Και αρχή της συζητήσεως ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, που έγινε επισήμανση κάποιων θεμάτων που μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερως αυτή τη στιγμή. Θέλω να στραφώ προς κάποιες μορφές ομάδων συνεργασίας μεταξύ κρατών. Μία μορφή είναι των μακροπεριφερειακών στρατηγικών που έχουν υπησέλθει, επευλήθησαν ούτως υπήν στη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως από κάποιες ομάδες χωρών που είχαν παράδοση και ανάγκη συντονισμού των πολιτικών τους για κάποια θέματα. Γεννήθηκαν γύρω από το νερό. Η πιο πρόσφατη δημιουργήθηκε γύρω από τις Άλπεις Παραδοσιακές περιοχές συνεργασίας όμως εκινήθηκαν και ο τρόπος. Από πάντοτε χώρες και κυρίως τοπικές και περιφερειακές κοινότητες συνεργάζονται για την επίλυση κοινών προβλημάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δέχτηκε αυτή την πρόκληση με την αρχή της ε, δαφικής περιφερειακής συνεργασίας στις συνθήκες ε, δικαιολογία αυτού του της συνεργασίες. Έπαιξε ένα ρόλο προπρογραμματισμού, συντονισμού, προϋπολογισμού κλπ. Δεν εξέτασε το θέμα όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση του καθεστώτος που έχουν αυτές τις συνεργασίες εντός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. μία αρχή διέπει αυτές τις συνεργασίες. Η δημοκρατική εκπροσώπηση των κοινοβουλευτικών του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου που εκπροσωπούν δημοκρατικώς οι φορείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εντός αυτών των μορφωμάτων δεν υπησέρχεται σε αυτές τις συνεργασίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω διευκολύνσεων και προγραμμάτων υπησέρχεται. Αλλά είναι ότι των δομών λήψεως αποφάσεων και που χρησιμοποιούν ευρωπαϊκούς πόρους και χρησιμοποιούν ευρωπαϊκές διευκολύνσεις, ακόμα και αν συμμετέχουν χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως, δεν μπαίνουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Σε αυτές τις ομαδοποιήσεις, σε αυτά τα μορφώματα, που δεν είναι κάτι ευκταίο, αλλά τελικά τα εκτιμούμε τις συνεργασίες, διότι πάντα έχει σημασία συνεργασία γειτόνων. Οι πόλεμοι δημιουργούνται μεταξύ γειτών στο κάτω-κάτω. Το ξεπέρασμα των συνόρων. Το ξεπέρασμα εντάσσεων παλαιών και προβλημάτων είναι κάτι σημαντικό. Είναι χρήσιμε οι συνεργασίε αυτέ και αυτά τα μορφώματα. Πώ μπορούν να ενταχθούν και να αφομοιωθούν, ούτω ώστε να υπάρχει καλύτερο δημοκρατικό έλεγχο και να μην περιοριζόμαστε σε γνωμοδότηση μέσω μια εκθέσεω κλπ. Δεύτερο ερώτημα συμμεριζόμενοι αυτά που είπε η κυρία Εμπερές και άλλοι για την Ευρωζώνη. Άλλη μια ερώτηση. Πώς ακριβώς θα ασκείται το δημοκρατικός έλεγχος. Ένας προϋπολογισμός ή ένα κονδύλι του προϋπολογισμού που είναι μια υπόθεση. Προς τα εκεί κινούμεθα περισσότερο. όχι προπολογισμό, κονδύλι για την Ευρωζώνη. Αν γίνει αυτό, τίθεται εκ νέου το πρόβλημα του τρόπου του δημοκρατικού ελέγχου πλευρά Κοινοβουλίου. Μέχρι τώρα, υπενθύμησε η κυρία Μπερέ, ξεπεράστηκε αυτό μέσω τη σπουδαία για το Κοινοβούλιο τη Ευρωζώνη και του Βασικού Κοινοβουλίου. Προσπαθήσαμε να συζητήσουμε το θέμα με τον συνάδελφο Μπροκ. Μεγάλες οι δυσκολίες υπήρξαν όμω. Η Επιτροπή ΕΚΟΝ μαζί με την Επιτροπή Προπολογισμών θα αξιολογούν το κονδύλι αυτό του προπολογισμού για την Ευρωζώνη. Θα συζητούνται διάφορες αλλαγές και τροποποίησεις. Η ψηφοφορία θα γίνεται με μόνη συμμετοχή των εκπροσώπων των χωρών της Ευρωζώνης. Και στο τέλος το Ευρωκοινοβούλιο θα δέχεται ή δεν θα αποδέχεται τα αποτελέσματα. Αυτή είναι μια δυνατότητα. Το πρόβλημα του δημοκρατικού ελέγχου, όχι μόνο πλευρά των κρατών, γιατί διατίθεται από τι χώρε του μέσω του προπολογισμού. Αλλά χρειάζεται δημοκρατικό έλεγχο χρήση ενό κονδυλίου ε, που διατίθεται για την Ευρωζώνη. Τίθεται αυτό σαν θέμα. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο που να μην οδηγεί σε διακρίσεις καμίας χώρας, ούτε, και ούτε κατά εκείνο που συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων διότι αποφασίζει το ECOFIN στο Συμβούλιο και όχι μόνο το Eurogroup. Φαίνονται όμορφα αυτά τα πράγματα αρχικά, αλλά υπάρχει κίνδυνος αποκλεισμός της δημοκρατικής εκπροσώπησης. Για το Βίζεγκραντ, συμμεριζόμενοι τις προηγηθήσεις παρατηρήσεις. Ερώτηση. Κύριε Ζήλερ, είναι δυνατόν να υπάρχει παραβίαση των αρχών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως εάν γίνεται, δημιουργείται αυτή η ομάδα για να αντισταθεί σαφώς στι αποφάσει Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Αυτό είναι σαφέ γιατί είναι δηλώσει σαφή κατά των αποφάσεων τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Εμποδίζονται συνεργασία μεταξύ κρατών μέλων. Τι μέσα μπορεί να χρησιμοποιηθούν για επιβολή κυρώσεων, για να αντιμετωπιστούν αυτές οι συμπεριφορές. άλλο συντονισμό των δράσεων και άλλο συντονισμό δράσεων με τελικό σκοπό την παραβίαση αποφάσεων τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Thank you, Ramon. Ευχαριστώ πολύ, ο Ραμόν Χαουράκη. Eh, λοιπόν, να σα ευχαριστήσω όλου. Θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η ιστορική εξέλιξη των υποομάδων αυτών ε, αυξάνονται, μειώνονται, ποια είναι η τάση. Γιατί από αυτά που μας είπατε ε, υπάρχουν δύο ζητήματα, δύο σημεία σύγχυσης τα οποία πρέπει να προσέξουμε. Πρώτον, ένα πράγμα είναι οι υποομάδες χωρών, ε, δαφικά συμφέροντα ας πούμε, που συνασπίζονται και άλλο πράγμα είναι η ενισχυμένη συνεργασία. Η ενισχυμένη συνεργασία ενοποιεί πολιτικές, ενώνει πολιτικές, πολιτικούς στόχους που μια σειρά από χώρε στα πλαίσια της Ένωσης θέλουν να διενεργήσουν, να πραγματοποιήσουν. Με ανησυχεί λοιπόν που είναι ενισχυμένη συνεργασία θεωρείται ως ε, ένα εργαλείο των υποομάδων χωρών. Όχι. Έχει, συγκεκριμένο μηχανισμό. Έχει συγκεκριμένους μηχανισμούς ε, η ενισχυμένη συνεργασία. Ε, υπάρχουν τρεις κατηγορίες, τις εξήγησε ο καθηγητής προηγουμένως. Έχει να κάνει όμως με στόχους της Ένωσης. Ενώ οι υποομάδες χωρών εκπροσωπούν το συμφέρον αυτών των χωρών. Επίση, αυτέ οι υποομάδες δεν πρέπει να τις συγχαίουμε με τις περιφερειακές πολιτικές ή με τις διασυνοριακές πολιτικές που ήδη διενεργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και εκπονεί και που τις επιτρέπει και που τις ενθαρρύνει, όπως είπε η κυρία Μπρέσο για τις Άλπεις. Ε, υπάρχουν πολλές περιφερειακές πολιτικέ που ενοποιούν αυτέ τι πολιτικέ. Ε, δεν είναι όμω υποομάδα χωρών αυτό. εδώ μιλάμε για ένα εθνικό μέτωπο εντό τη Ένωση και αυτό είναι που με απασχολεί περισσότερο ε, με τι υποομάδε χωρών. Διότι σε πολλέ περιπτώσει ο στόχο αυτών των υποομάδων είναι να. Το αποτέλεσμα είναι να ανοίγουν τα χάσματα ακόμα περισσότερο. Και αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο μεγάλε ρογμέ Σε οικονομικό επίπεδο βορράς-νότος όλο και περισσότερο τα τελευταία δέκα χρόνια και Ανατολή, Δύση για τη μεταναστευτική πολιτική κτλ. Το να προσθέτουμε νέε ρογμέ στην ευρωπαϊκό οικοδόμημα είναι εξαιρετικά ανησυχητικό κατά τη γνώμη μου. Εξού λοιπόν και η αρχική μου, το αρχικό μου ερώτημα, η εξέλιξη αυτών των υποομάδων, ποια είναι, ποιε είναι οι τάσει υπάρχει αύξηση ή μείωση. ο καθηγητή μακάλι που έκανε και μια πολιτική περιγραφή αυτών των ομάδων να μπορεί να μα πει κάτι ενδεχομένω. Και δεύτερο ερώτημα, θα πρέπει να περιορίσουμε περισσότερο τη δυνατότητα ή εν πάση τις απαγορεύσεις που προβλέπονται για αυτές τις υποομάδες ε, διότι όλο και πιο συχνά αποτελούν εμπόδιο στη δράση τη Ένωση. Η Ευρώπη διαπραγματεύεται αυτή τη στιγμή μια συμφωνία με τι χώρε του Μερκοσούρ, παραδείγματο χάρη, με την Αργεντινή, τη Βραζιλία κτλ. Είναι πιθανό ε, μια σειρά από χώρε που ε, παράγουν κρέα, ε, παράγουν σιτάρι, να διαφωνήσουν, να φτιάξουν μια υπομάδα και να συνασπιστούν. Και ποιοι για άλλα τέτοια. Να μην υπάρχει, λοιπόν, να μην υπάρχουν περισσότερα εμπόδια. Ευχαριστώ. Ο Τζόρτ Σέφιλ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και τους εμπειρογνώμονες. Να επανέλθω λίγο σε αυτά που είπε η κυρία Μπρέσο και η κυρία Σπινέλη. Ίσως ξεχάσετε αυτό το κομμάτι της ιστορίας. Το Βίσεγκρα δημιουργήθηκε το 1991 και η Ευρωπαϊκή Ένωση το καλωσόρισε, γιατί ήταν ένδειξη της ετοιμότητας των κρατών αυτών να εισέλθουν σε μια ε, διαδικασία συνεργασίας. Και αν πάτε και ακόμα πιο πίσω στην ιστορία, θα δείτε ότι αυτή η περιοχή είχε χαρακτηριστεί από έντονες ε, διαμάχες ανάμεσα στις χώρες εκείνες. Γι' αυτό λοιπόν το V4 είναι μία ε, περίπτωση success story στην Ευρώπη. Τώρα αν το θέλουμε ή όχι είναι άλλο πράγμα. Έπειτα, ε, το, η V4 είναι μόνο τέσσερις από τις 11 πρώην κομμουνιστικές χώρες που ανήκουν τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με άλλα λόγια δηλαδή, πρέπει να δοθούν κάποιες εξηγήσει ε, και να δούμε γιατί είναι τέσσερα μέλη και όχι 11. Αν ανατρέξουμε ιστορικά θα βρούμε διάφορα, αλλά θα δούμε επίσης και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση των 15 ε, ποτέ δεν συμφιλιώθηκε με το κομμουνιστικό παρελθόν της Ευρώπης. Δεν θα μπω βέβαια σε λεπτομέρειες. Αλλά με λίγα λόγια, αυτό το κομμάτι της ευρωπαϊκής ιστορίας ποτέ δεν αναγνωρίστηκε επίσημα δεν αποτελεί μέλος του αφηγήματο. Και ξέρετε, πολλοί από τους ε, υπεύθυνου, πολλοί από αυτούς που δολοφόνησαν Ούγκρους μετά την ε, Επανάσταση του 1954 ζουν ακόμα. Υπάρχουν ουσιαστικές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που κανείς δεν έχει ασχοληθεί με αυτά. Έπειτα, ένα κομμάτι της ιστορίας των 11 ε, χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν ότι αυτές οι χώρες ποτέ δεν είχαν απικιακό ε, παρελθόν, δεν είχαν απικιοκρατικό μάλλον παρελθόν. Ήταν αντίθετα απικίες. Η δική μου χώρα, η Ουγγαρία, ήταν κομμάτι τριών αυτοκρατοριών, της Οθωμανικής, της ε, Αυστριακής και της Σοβιετικής. Και δεν είναι ευχάριστο να ξέρεις ότι ανήκεις, ε, ότι έχεις ένα τέτοιο παρελθόν μάλλον. Αυτό που λείπει είναι μία σχέση ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 15-14 μάλλον και σε εκείνη των 11 είναι μία σχέση ισότητας στην οποία μάλιστα είχαν στηριχθεί και οι πατέρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπάρχει αυτό το αίσθημα. Και αυτές οι χώρες ποτέ δεν ε, λήφθησαν ε, στα σοβαρά. Γι' αυτό, ναι, ένα παράδειγμα, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση διαπραγματεύεται με, την Αλτική, με τη Λατινική Αμερική, είναι αδιανόητο να λείπει η Ισπανία από τις διαπραγματεύσεις. Όταν ε, διαπραγματεύεται με τη Ρωσία, είναι αδιανόητο να λείπει η Πολωνία. Και αυτό για μένα είναι μια έλλειψη που δεν αντιμετωπίστηκε ποτέ. Δεν υπάρχει δηλαδή θεώρηση των χωρών αυτών ως ίσες. Και κρύβονται και κάποιες παγίδες πίσω από αυτό επίσης, παγίδες οι οποίες έχουν κοινωνικό, οικονομικό υπόβαθρο. Και υποπτεύομαι ότι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ξανά έκανε στον εαυτό της την ερώτηση του τι είναι μετά τη διεύρυνση του 2014 και 2017. Με άλλα λόγια, η επικουρικότητα που θα έπρεπε να είναι αναπόσπαστο κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει εφαρμοστεί στις 11 χώρες αυτές. Τώρα γίνεται παράκαμψη των αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, να δούμε τι γίνεται με το δικαστήριο και με τον πίνακα επιδόσεων της Κομισιόν. Θα δείτε λοιπόν, αν κοιτάξετε σε αυτό τον πίνακα, ότι αυτές οι δέκα χώρες δεν έχουν άσχημα αποτελέσματα. Αντίθετα, η Ιταλία έχει άσχημες επιδόσεις. Κανείς όμως δεν ανησυχεί γι' αυτό. Ανησυχούν για την Ουγγαρία, την Πολωνία, τη Ρουμανία και τις υπόλοιπες χώρες. Αν δούμε τις διαδικασίες επί παραβάση, Αυτές οι χώρε δεν είναι στην κορυφή του καταλόγου. Η Ισπανία, από την άλλη, δεν τα πάει και τόσο καλά. Ε, τα μέσα ενημέρωση βέβαια έχουν διαφορετική άποψη, αλλά δεν νομοθετούν αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ε, μπορείτε να επιλέξετε, αγαπητοί προσκεκλημένοι, ποιος από εσά θα αρχίσει πρώτος. Οι κυρία προηγούνται. Ευχαριστώ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσες οι ερωτήσεις σας. Θα αφήσω στον κύριο Τσίλερ να απαντήσει τα νομικά ερωτήματα ε, και να σταθώ λίγο στην ομάδα του Βίσεγκραντ και στις γενικότερες ερωτήσεις ε, που αναφέρονται στις υποπεριφερειακές ομάδες και στο αν θα έπρεπε να υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί για τη δημιουργία τέτοιων ομάδων στο μέλλον. Ένα επιχείρημα, μάλλον κάτι που παρατήρησα, μια διαφορά ανάμεσα σε όλες τις παρεμβάσεις είναι οι διαφορετικές αντιλήψεις για την ε, συνεργασία, για την περιφερειακή συνεργασία. Αυτό οφείλεται σε διαφορετικές ερμηνείες ή διαφορετικές επιθυμίες για από τη μία μελλοντικές διευρύνσεις και για τις διευρύνσεις που έχουν ήδη γίνει στο παρελθόν. Και εδώ επιστρέφουμε στο ερώτημα του ποιες είναι οι κοινέ ευρωπαϊκές αξίες και ποια είναι τα θεμέλια της Ένωσης σήμερα. Έχω την εντύπωση πως υπάρχει αυξανόμενη δυσαρέσκεια ε, για αυτήν την εξάρτηση από την κατεύθυνση που παίρνει η Ευρώπη. και συμφωνώ πως δεν πρέπει να συγχύουμε την ενισχυμένη συνεργασία και τις ε, υποπεριφερειακές ομάδες όσο δυνατές και να είναι αυτές. Αλλά ε, η ιδέα ότι ο γαλλογερμανικός άξονας ή η Γερμανία θα πρέπει να αποκτήσουν έτσι ενισχυμένες ε, δυνάμεις είναι κάτι το οποίο έχει επιπτώσει στην ευρωπαϊκή πολιτική. τα μικρότερα κρατημέλη, ανεξάρτητα από το αν είναι του Νότου, της Ανατολής, ε, έχουν κάποιες δυσκολίες με αυτό. Όμως μην ξεχνάμε ότι υπάρχει το Κοινοβούλιο, υπάρχει το Συμβούλιο. Είναι ε, πάρα πολύ μεγάλη γενίκευση να πούμε ότι η Γαλλία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν τα ενία. Είναι όμως πολιτική η πρόκληση, την οποία δεν μπορούμε να λύσουμε με τα όργανα που έχουμε. Γι' αυτό λοιπόν συμπεραίνω πως θα έπρεπε ίσως να γίνει πιο εύκολο στο μέλλον να αποτρέπονται ε, τέτοιες ε, ομάδες, να μην επιτρέπουμε τη δημιουργία τους, να τις αποθαρρύνουμε και να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που έχουν δημιουργηθεί. Από την άλλη, θα σας τα πούν και οι συνάδελφοι καλύτερα, οι ποσοστώσεις μετεγκατάστασης αναφέρθηκαν. Αναφέρθηκε και η απόφαση του δικαστηρίου μετά την ε, ένσταση που υπέβαλε η Ουγγαρία και η Σλοβακία. Υπάρχουν λοιπόν τα νομικά μέσα για να λύσουμε αυτά τα προβλήματα. Δεν χρειάζεται να δημιουργήσουμε νέους κανονισμούς. Τώρα, εάν και κατά πόσο θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να εφαρμόσει αυτούς τους κανόνες είναι το ζητούμενο, είναι το καυτό θέμα. Υπάρχουν κάποια θέματα που έχουν μεγαλύτερη ορατότητα από την άλλη. Είπα και στην αρχή ότι υπάρχουν πολλοί τομείς όπου λάθος εντοπίσαμε προβλήματα. Πρέπει λοιπόν να δούμε τι γίνεται με, την, με, με, τα, με τους προβληματικούς τομείς, με την κατάσταση των προσφύγων, να αποφύγουμε τις γενικεύσεις. Είναι μια μεγάλη κρίση που διανύουμε αυτή τη στιγμή, σίγουρα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Καταλαβαίνω πως υπάρχουν πολλές ανησυχίες στις χώρες αυτές. Βέβαια, υπάρχουν και άλλες χώρες που έχουν ανησυχίε για άλλα θέματα και χώρε χώρες του Νότου, ας πούμε, έχουν σοβαρέ ανησυχίε γι' αυτό. Το γεγονός ότι υπάρχει τέτοια πολυμορφία στην Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Ένωση καλύπτει τέτοια μεγάλη γεωγραφική έκταση ε, είναι κάτι που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Οι βόρειες χώρες ε, έχουν ανησυχίες ε, από την πλευρά της Ρωσίας. Είναι λοιπόν πολιτική θα έλεγα η πρόκληση και όχι τόσο νομική. Μετά ε, έγινε η ερώτηση αν υπάρχει έτσι ιστορικά η τάση να δημιουργούνται τέτοιες υποομάδες. Υπάρχουν διάφορες τάσεις. Ακούσαμε και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στήριξε αυτές τις ομάδες στην αρχή για τη διασυνοριακή συνεργασία, για τη στάση του στο ΝΑΤΟ, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ενθάρρυνε αυτήν την περιφερειακή προσέγγιση για να απορροφηθούν και πιο γρήγορα πόροι. Να πω τώρα εδώ ότι υπήρχαν και διάφορες επομάδες στην νότιο-ανατολική Ευρώπη, οι οποίες διαλύθηκαν πολύ γρήγορα μόλις επέτυχαν το στόχο τους, να γίνουν δηλαδή μέλη του ΝΑΤΟ. Μετά ε, υπήρχαν επίσης διάφορες ομάδες που διαλύθηκαν μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου. Θα έλεγα λοιπόν πως δεν υπάρχει κάποια γενική τάση για ενίσχυση της ε, υποπεριφερειακής συνεργασίας, αλλά πρέπει να γίνει και ένας διαχωρισμός ανάμεσα στις λειτουργικές ομάδες, οι οποίες δεν σχετίζονται με γεω... δεν, δεν έχουν γεωγραφικά μάλλον κριτήρια και τις άλλες. Δεν ξέρω αν έχουμε άλλο χρόνο, αλλά αν υπάρχει και άλλο χρόνο μπορούμε να κάνουμε και ένα δεύτερο γύρο απαντήσεων, αν θέλετε. Ευχαριστώ πολύ. Πολλές ερωτήσεις για να μπορέσω να απαντήσω σε όλες. Δεν έχω και τις απαντήσεις άλλωστε σε όλες. Κατανοώ το βασικό ερώτημα κάποιες ομάδες θα μπορούσαν να αντιταχθούν στο ευρωπαϊκό κύρος και στην ομοιογένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ομάδα του Βίζεγκρατ μας έρχεται στο νου κυρίως. Δεν συμμερίζομαι αυτή την προσέγγιση. Από πλευρά νομικής, όπως εξηγήθηκε, υπάρχουν όρια συγκεκριμένα και αυτή η ομοιογένεια δεν προσωπείται για όλα τα ζητήματα. Αν πάτε αυτές τις τέσσερις για λόγους πολιτικής απόχρωση Κάποιε ανήκουν στην Ευρωζώνη, κάποιε όλε και υπάρχουν διαφορετικέ προοπτικέ. Το καλοκαίρι είδατε πολλά μηνύματα που έδειχναν διαφωνία εντός αυτού του μορφώματος της ομάδας των χωρών Βίζεγκραντ. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν μιλάμε για ομάδες. Μην αρχίσουμε να θεωρούμε ότι όσον αφορά τα θέματα και τι πολιτικέ έχουν ομοιογένεια. Δεύτερο, ο κίνδυνος. Να συγκεντρωθούμε επί κάποιων κακών μαθητών της τάξης. Το θέμα είναι η διαδικασία επί παραβάση. Είναι ιδιαίτερη διαδικασία. Αυτό που φυζητείται σε κάποιες χώρες όσον αφορά την εφαρμογή του κράτους δικαίου και των αξιών συγκρίνεται με όλα τα κράτη-μέλη τα οποία, κατά των οποίων κινείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δικαστικά. Όπως διαφοροποιήσει όσον αφορά τους γενετικά τροπημένους οργανισμούς. Υπάρχουν διαφορετικού είδους προσφυγές στο δικαστήριο. Παρόλο που όλες είναι νόμιες προσφυγές, δημοκρατικός έλεγχος, περίπλοκο θέμα. Δεν υπάρχουν παντού ε, ήδη δημοκρατικοί έλεγχοι για το μέλλον, για την Ευρωζώνη. Ο προπολογισμό της, μηχανικός πώς θα διαρθρωθεί μέσω ε, του δημοκρατικού ελέγχου πρέπει να είναι ισχυρότερο. στο μέλλον. Υπάρχει μία δράση, αντίδραση, χρειάζεται χρόνος για την αντίδραση. Αν υπάρχει προπολογισμό για την Ευρωζώνη, και πέρα από το κονδύλι του κοινού προϋπολογισμού θα υπάρχει και ανάγκη ε, συγκεκριμένου φορέα, κυρίως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που θα πρέπει να ασχολείται με τον έλεγχο. Τώρα, αν πρέπει να υπάρχει νομικός περιορισμός της συνεργασίας περιφερειακής, ad hoc, ενισχυμένης συνεργασίας, εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν εργαλεία ελέγχου είναι αρκετά ισχυρά. Πρέπει να έχουν πιο μεγάλη θέση στη δημόσια συζήτηση στην Ευρώπη, δεν γνωρίζω. Γίνονται συζητήσεις στο Ευρωκοινοβούλιο. Χρειάζεται στενότερη επαφή με τις υποομάδες. Υπάρχουν οι εκπρόσωποι των περιοχών και των περιφερειών και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν χρειάζεται ξεχωριστό φορέας. συμμερίζομαι εν γέννη τα υποθέντα από τους δύο προλαλήσαντες. Όσον αφορά τις εξελίξεις, δεν διαπιστώνουμε αύξηση των υπομάδων, αντιθέτως μάλιστα. Δεν υπάρχουν ιβυρικές υπομάδες, Φερρυπίν, λατινικές υπομάδες, παρά κάποια ευχολόγια που έχουν ακουστεί. Όπως υπόθηκε σωστά, η συζήτηση εστιάζεται επί της ομάδας Βίζεγκρατ και υπάρχει σύγχυση μεταξύ της ομάδας του Βίζεγκρατ και των πιο συγκεκριμένων θέσεων της κυβερνήσεως της παρούσης της Πολωνίας, παρούσης λέγω, και της παρούσης ουγγρικής κυβερνήσεως. Με αλλαγέ μέσω εκλογών μπορεί να αλλάξει τα πράγματα. Έτσι γίνει και στο παρελθόν. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να το έχουμε υπόψη παραβιάσεις του δικαίου. Το πρόβλημα δεν είναι το περιεχόμενο των συνθήκων, αλλά ποιες οι κυρώσει και ποιος μπορεί να τις ξεκινήσει, να τις εφαρμόσει τις κυρώσεις. Το άρθρο 7, όπου το Κοινοβούλιο μπορεί να κάνει κάτι. Η διαδικασία επί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να κινήσει κάτι τέτοιο. Υπάρχουν πολιτικές επιλογές. Ξέρετε καλύτερα από μένα ότι στο Κοινοβούλιο οι αποφάσει εξατώνται από την ύπαρξη πλειοψηφία και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανάλογα από την συνετή προσέγγιση που ακολουθεί ανάλογα με τη χρονική στιγμή. Τώρα σε πιο σημαντικά ουσιαστικά ζητήματα, η Ευρωζώνη και η δημοκρατική εκπροσώπηση. πρέπει να γίνεται διάκριση μέσω των συνθηκών του ισχύοντο ε, δικαίου και μελλοντικών εξελίξεων. Σε μελλοντικέ εξελίξει, μόνο οι πολιτικέ δυνάμει στα κράτη-μέλη θα επιτρέψουν, δεν θα επιτρέψουν ένα κοινοβούλιο της Ευρωζώνης ή να ασχολείται το Ευρωκοινοβούλιο με τον προϋπολογισμό της Ευρωζώνης που θα ψηφίζεται από την Ολομέλεια πρέπει να επιμείνουμε επί της συγχύσεως του πολιτικού λόγου και τι γράφεται στα ΜΜΕ όσον αφορά την Ευρωζώνη που είναι η Ευρωζώνη των 19 και την Ευρωζώνη που θα μπορούσε να φτάσει μέχρι 27 χώρες μέλη. Αν η Δανία αλλάξει γνώμη, παραδείγματος χάρη, ίσως θα διοργανώσει ένα νέο δημοψήφισμα. Η Δανία το ίδιο ισχύει για τη Σουηδία. Αν αλλάξουν εκλογή άποψη, θα διεξαχθεί νέο δημοψήφισμα για τη συμμετοχή της Σουηδίας στο Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα. Πρέπει να έχουμε υπόψη λοιπόν ότι συνδέοντας τα δύο μπορούμε να πούμε ή τα κάνουμε όλα μαζί με τις παρούσες χώρες της Ευρωζώνης και χωρίς τις άλλες θα είναι δύσκολα τα πράγματα αντί αυτή η περίπτωση. Υπάρχει υποχρέωση ανοίγματο πάντα και για την Ευρωζώνη. Τα κράτη-μέλη που επιθυμούν θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια για να ενταχθούν. Αν πληρούν τα κριτήρια και δεν το θέλουν, λυπούμε, θα υποχρεωθούν. Πώ δεν ξέρω. Είναι κάτι που δεν το τονίζουμε αρκετά και είναι μια απάντηση που θεωρώ σημαντικότατη. Τα κράτη-μέλη που ανησυχούν, οι κυβερνήσει των κρατών μελών που ανησυχούν, που δεν συμμετέχουν στην Ευρωζώνη, Κάντε λοιπόν τα αναγκαία για να μπείτε. Η νομική και πολιτική απάντηση είναι αλληλένδετες σε αυτό το τομέα. Το fiscal compact, όπως λέμε στη γλώσσα των Βρυξελών και όχι μόνο. Για την ώρα έχουμε χρόνο μέχρι αρχές του επομένου έτους. Δεν είδα πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ούτως ώστε το fiscal compact να ενταχθεί στο παράγωγο δίκαιο. Ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτε το Ευρωκοινοβούλιο δεν δεσμεύονται από αυτά που έχουν συμφωνήσει κάτι μέλη μεταξύ τους σε μία συνθήκη. Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όλος ιδιαίτερος, αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έρχεται με προτάσεις μπορεί να πει ναι, αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι. Επειδή υπάρχει ένα άρθρο στη συνθήκη τη λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω το λέει αυτό, όχι. Τα κράτη-μέλη υποχρεώνονται να ζητήσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το κάνει αυτό. Μικρή προσε... Ε, διευκρίνηση. Το πρόβλημα της συμφωνίας του Ιπρούμ προέβλεπε το ίδιο πράγμα. Όμως, εξακρίβωσα πρόσφατα ότι υπάρχουν κάποια άρθρα της συμφωνίας του Πρίμ που δεν μεταφέρθηκαν στο παράγωγο, όπως ε, υπάρχουν σε συμβάσει μεταξύ κρατών μελών. Το δίκαιο έχει τα όρια του. Έχουμε λοιπόν την Ευρωζώνη των 19 ή και θα μείνει έτσι ή θέλουμε μια ευρωζώνη που θα καλύπτει όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δημοκρατική εκπροσώπηση μετά. Με μεταρρύθμιση των συνθήκων μπορούμε να προβλέψουμε τα πάντα. Για την ώρα όμως δεν υπάρχει μεταρρύθμιση των συνθήκων που λαμβάνει η χώρα. Καλύτερα από μένα ξέρετε τις λεπτομέρειες. Το περιθώριο το ελιγμών είναι στα χέρια του Ευρωκοινοβουλίου. Έχουν δημιουργηθεί διακοινοβουλευτικές ομάδες στο Ευρωκοινοβούλιο που μπορούν να πούν λέγοντας ότι συνεδριάζουμε, κάνουμε μια πρόταση, δεν μπορούμε προφανώς να περιορίσουμε την ολομέλεια να ακολουθήσει όμως. Αυτοί που δεν θα είναι στη διακοινοβουλευτική ομάδα θα έχουν την τάση να κινηθούν αντίθετα. Αυτή εδώ η Επιτροπή μας έχει τα μέσα να φανταστεί κάποιες λύσεις κάποια στοιχεία γεννήσης κάποιων δομών σε όλη την προπαρασκευαστική φάση του προπολογισμού. Και σαν ελεγκτές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να υπενθυμίσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι κάποτε δημιουργούσε ομάδες κρούσης, task force, που ασχολούνταν με συγκεκριμένα θέματα. Είχα ασχοληθεί πολύ τότε με τις task force για τις τα υπερπόντια διαμερίσματα, κάτι που εξαφανίστηκε. Τώρα η DG Regio, η Γενική Διεύθυνση Regio για τι διεθνεί σχέσει ασχολείται με αυτά. Το Ευρωκοινοβούλιο μπορεί να σπρώξει, να πιέσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διοργανωθεί καλύτερα για να λάβει υπόψη και τι λειτουργικέ ομαδοποίησει και τι γεωγραφικέ. Καμιά φορά ε, είναι γεωγραφική φύσεω οι λειτουργικέ υποομάδε. Ε, και βέβαια καθορίζονται αυτέ οι υποομάδε από τη γεωγραφία. Είναι λογικό αυτό. Thank you very much. Ευχαριστώ, σας ευχαριστώ και για τις ιδέες ε, που ε, μοιραστήκατε μαζί μας. Ε, δεν ολοκληρώνουμε βέβαια τη συζήτηση αυτή. Μόλις ξεκίνησε. Θα συνεχιστεί σίγουρα τα επόμενα χρόνια και διαπιστώνω από όλα αυτά που μας είπατε ότι είναι δύσκολο ακόμα και να ορίσουμε το φαινόμενο αυτό. Διότι ο καθένα το προσεγγίζει από διαφορετική σκοπιά. Χαίρομαι πάντω ιδιαίτερα που εσεί ε, το καλύψατε από διάφορε πτυχέ. Ελπίζω να μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση. Για την ώρα ευχαριστώ ιδιαίτερω για τη συνεισφορά σα. Σας ευχαριστώ όλους για τις παρεμβάσεις σας. Λοιπόν, σε δύο λεπτά ψηφίζουμε. Ας περιμένουμε να έρθουν και οι υπόλοιποι. Uh, yeah. Oh, so I'll be looking at you all the time, okay.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 <clears throat> Αγαπητοί συνάδελφοι, ας κάνουμε έναν έλεγχο για να δούμε αν λειτουργούν οι κάρτες και τα μηχανήματα. Άρχεται η ψηφοφορία. Α, ah, where is the opening of... Ας αρχίσουμε λοιπόν τη δοκιμαστική ψηφοφορία ελέγξτε τις κάρτες σας και ψηφίστε παρακαλώ. Δεν έχουν ελέγξει όλοι οι συνάδελφοι αν λειτουργούν τα μηχανήματά τους. Δύο Συνάδελφοι δεν έχουν ψηφίσει. Είστε σίγουροι ότι λειτουργεί, εντάξει. Περβάνησε δεν έχει κάρτα. Είναι κάποιος άλλος που έχει ξεχάσει την κάρτα. Να φωνάζετε λοιπόν για να σας μετρήσουμε. Μόνο μία ψηφοφορία έχουμε σήμερα. Ας αρχίσουμε λοιπόν Ψηφίζουμε το σχέδιο γνωμοδότησης για την έκθεση για την ε, θεγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2017. Συμβιβαστική τροπολογία 1. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Θα μας πάρει λίγο περισσότερο χρόνο γιατί είναι δύσκολο να δούμε, είναι στα γράμματα περίεργα. Τροπολογία 7, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 8. Προστίκη. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος στην τροπολογία 8. Άρχεται η ψηφοφορία. Ένας παραπάνω από το ΕΛΚ. Φροντίστε το. Ψεφίσατε όλοι. Απορρίπτεται. Ε, συγγνώμη γιατί δεν βλέπω. Έχω το φως από πίσω μου. Όλα εναντίον μας είναι. Απορρίπτεται. Τροπολογία 9. Υπέρ. Κατά. Έλεγχο στην 11. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 8 ψήφοι υπέρ, 10 κατά. Παρεμβάνω δεν αλλάζει κάτι. Δεν θα επηρεάσει λοιπόν το αποτέλεσμα. Λυπάμαι που στο λέω. 14. Υπέρ. Απορρίφθηκε η προηγούμενη. Okay, are you, can we go on? Μπορούμε να συνεχίσουμε. Τροπολογία 14. Υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά την τροπολογία 14. Ένα one e too much again. Again, e Ένας παραπάνω από το ΕΛΚ ξανά. Εντάξει τώρα. Απορρίπτεται. 11 ψήφοι κατά. Τροπολογία 15 υπέρ, κατά, ας ελέγξουμε. Νομίζω πως εγκρίνεται, αλλά ας ελέγξουμε. Πέρας, απορρίπτεται. Τροπολογία 16. Υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε πάλι. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 17 υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε πάλι. Τροπολογία 17. Υπερβάνης ψηφίζεις υπέρ, 10 προς 10 απορρίπτεται. Συμβαστική 3, ποιος είναι υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 24, υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 25, υπέρ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Εγκρίνεται, συγγνώμη, εγκρίνεται, λέει πρόεδρος. Τροπολογία 26, προφορική τροπολογία από την Μπάρμπαρα. Υπάρχει κάποια ένσταση, όχι. Ψηφίζουμε λοιπόν, περ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 29. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τριάντα. Υπέρ. Κατά. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. The vote is closed. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 31. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 41 υπέρ κατά. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά τη 41, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Περνάμε στην τελική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ονομαστική κλίση. Πέρας. 15 υπέρ, 5 κατά. Yeah, but uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε συνάντηση των συντονιστών στις 2.30 και 3.30 η Επιτροπή. Σας ευχαριστώ.